Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Να ξεκινήσει η συνεδρίαση, να καλωσορίσω αυτούς που είναι ήδη εδώ και θα ήθελα να περάσω στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Σας διανεμήθηκε την ε, Πέμπτη, είχατε την τελική εκδοχή. Να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα το πρωί με πριν από τις συνεδρίες με τα Εθνικά Κοινοβούλια που θα ξεκινήσει στις 10, θα θέλαμε να συζητήσουμε δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη, η έκθεση του Ραμών Χαουρέγη για την ηλεκτρονική δημοκρατία και την ε, ε, γνωμοδότησή μου για το σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Επίσης, ε, θα ήθελα να σας πω ότι ο πρέσβης της Σλοβακικής Προεδρίας, ο Πέτερ Γιάβορτσικ, έχει έναν έκτακτο τριμερή διάλογο στις 10 και θα έρθει νωρίτερα, εάν υπάρχει δυνατότητα να ξεκινήσει λίγο νωρίτερα η συνεδρίαση με τα Εθνικά Κοινοβούλια και να του δώσουμε το λόγο στον πρέσβη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε πριν από τις 10. Εάν συμφωνείτε και έχουμε και αρκετά μέλη στην αίθουσα, θα του ζητήσουμε να λάβει το λόγο πριν από τις 10. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις για την ημερήσια διάταξη, και δεν θέλει κάποια τροποποίηση κανείς, θεωρώ ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη με τα σχόλια τα οποία σας ανέφερα. Σημείο 2. Ανακοινώσει της Προέδρου. Να σας ενημερώσω πολύ σύντομα ότι συμμετείχα στην συνεδρίαση της Ολομέλειας της Κόζακ στην Πρατισλάβα November Στι 15 Νοεμβρίου συζητήθηκαν δύο σημαντικά θέματα. Το ένα ήταν ο ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στη διαδικασία λήψη αποφάσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το άλλο ήταν η TTIP. Θα λάβατε την αναλυτική ε, έκθεση όταν θα συνταχθεί. Δεν θα σας καθυστερήσω λοιπόν ε, λέγοντάς σας ε, περισσότερες πληροφορίες. Ε, να πω απλώς ότι έγινε η συνεδρίαση, η συζήτηση ως συνήθως ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και νομίζω ότι ως Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γέφυρες με τα Εθνικά Κοινοβούλια και να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η γενικότερη αίσθηση όμως που έχω είναι ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια εξακολουθούν να διαπιστώνουν ότι υπάρχουν δυνατότητες ε, να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εξακολουθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μην συζητούμε αυτή τη σχέση με τα εθνικά θεσμικά όργανα, κυρίως με τις εθνικές κυβερνήσεις. Αυτή η πρόκληση λοιπόν να βρεθεί μια κοινή γλώσσα για το συνταγματικό ρόλο κάθε επίπεδου του Κοινοβουλίου και των κοινοβουλευτικών θεσμών εξακολουθεί να εκκρεμεί ε, στην ε, Ευρωπαϊκή συζήτηση. Οι επόμενε συνεδριάσει τη ΚΟΖΑΚ στη Μαλτέζικη Προεδρία θα γίνουν στη Βαλέτα στι 22 και 23 Ιανουαρίου, μόνο για του Προέδρου των Επιτροπών και στη συνέχεια 28 ε, με 30 Μαου για την Ολομέλεια της ΚΟΖΑΚ. Θα ήθελα να σας ζητήσω να προσπαθήσετε να πείσετε την πολιτική σας ομάδα ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος εκπρόσωπός σας στις συνεδριάσεις της ΚΟΖΑΚ. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πλατφόρμα και θα μπορούσε να είναι και πλατφόρμα επιρροής στις συζητήσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Να σας πω ότι στην τελευταία συνεδρίαση στην Πρατισλάβα συμμετείχα ως πρόεδρος της ΑΦΚΟ. Εξορισμού λοιπόν Είμαι ο αντιπρόεδρος της ε, αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Πρατισλάβα. Εκτός από μένα ήταν εκεί ο Μάρκος Πρέτσελ από το ΕΝΕΦ. E Αυτή ήταν δηλαδή η εκπροσώπηση της ε, ΚΟΖΑΚ, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μάλλον στην ΚΟΖΑΚ. Να περάσουμε στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης, συστάσεις των συντονιστών. Δεν έχω κάποια σύσταση σήμερα θα γίνει συνεδρία των συντονιστών την επόμενη εβδομάδα στις 5 Δεκεμβρίου. Θα σας ενημερώσω λοιπόν μετά. Να περάσουμε πέσως λοιπόν στην ηλεκτρονική δημοκρατία και στο Ραμόν Χαουρέγγι για να ξεκινήσει λοιπόν η συζήτηση. Ραμόν, να σου δώσω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Όπως θα θυμάστε, η γνωμοδότηση για την ηλεκτρονική δημοκρατία θέλει να προτείνει κάποιες συστάσεις στα πλαίσια της εξίσωσης δημοκρατία-τεχνολογία. Όπως θα θυμάστε, ε, αυτό που θέλω είναι να θέσω το πλαίσιο αυτής της συζήτησης. Ε, ξεκινάμε από την προϋπόθεση ότι η δημοκρατία, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, πάσχει αυτή τη στιγμή και πλήττεται από μια σειρά από επιθέσεις από την προπτική της γενικότερης δυσαρέσκειας καταρχάς των πολιτών, ε, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τους φορείς που λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις, ε, τη δυσαρέσκεια την οποία προκαλεί η κρίση, τους πολίτες, ε, την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους θεσμούς εν γέννη. Σε αυτή λοιπόν την ειλικρινή διαδικασία προβληματισμού και αυτοκριτικής που κάνουμε ε, όσον αφορά την κατάσταση της δημοκρατίας μας, προσπαθούμε να διερευνήσουμε τι μηχανισμούς μας προτείνουν οι τεχνολογίες της επικοινωνίας. Αυτή η νέα κοινωνία της πληροφορίας, ε, οι τεχνολογικές διακλαδώσεις εν γέννη προκειμένου να ε, βελτιωθεί η δημοκρατία. Όπως θα θυμάστε αυτό είναι το θέμα μας. Δεν ε, θα ήθελα να επαναλάβω το κείμενο της γνωμοδότησης. Απλώς, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επενθυμίσω ότι αυτές τις τελευταίες ημέρες ε, όταν ε, εξέπνευσε η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών, περίπου 230 τροπολογίες λάβαμε από τις διάφορες πολιτικές ομάδες και κατά την άποψή μου, επειδή τις μελέτες όλες είναι πολύ ενδιαφέρουσες, κάποιες συμπληρώνουν, κάποιες άλλες προσθέτουν κάποια πράγματα, Ε, κατά την άποψή μου θέτουν και θέματα υποχρεωτικού προβληματισμού. Ε, προσπαθώ να βρω κάποιες συμβιβαστικές λύσεις για τις περισσότερες από τις παραγράφους της γνωμοδότησης, αλλά πιστεύω ότι το καλύτερο θα ήταν, κυρία Πρόεδρε, να ακούσουμε ή δυνατόν, δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα σήμερα, ε, τους διάφορους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων, ώστε να μας εκθέσουν ε, υπό ποιο πνεύμα ε, υπέβαλαν τις τροπολογίες τους. Ε, αν μου επιτρέπετε κυρία Χούμπνερ, εγώ ε, θα απαντήσω στη συνέχεια, διότι θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η αίσθηση των τροπολογιών μας, γιατί η ουσία είναι να ακούσουμε τι έχουν να πούνε. Αν συμφωνείτε, η Πρόεδρος. Ναι, νομίζω λογικό είναι να γίνει αυτό. Να ξεκινήσουμε με το ΕΛΚ. Ο Τζορτ Σέπφλιν θα μιλήσει εξ ονόματος του Κρίστιαν Νταν Πρέντα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και βεβαίω δεν θέλω να ευχαριστήσω για τον Ισίδη για την προετοιμασία του. Ο κύριος Πρέντα μου ζήτησε να διαβάσω την εξή δήλωση, μιας και δεν μπορούσε να παρευρεθεί, για το ζήτημα της ηλεκτρονικής δημοκρατίας. Είχε ανακοινωθεί ε, ότι ο κύριος Πρέτα θα υποβάλει 16 τροπολογίες στην τελευταία μας συνάντηση. Άλλοι συνάδελφοι όπως ο κύριος Μακάλεστερ επίσης έχουν ε, υποβάλει τροπολογίες τις οποίες θεωρούμε χρήσιμες γιατί με επιδιώκουν να διευκρινίσουν ε, σημεία του κειμένου. Ένα κείμενο που ήδη βέβαια είναι πολύ καλό. Έχουν συνολικά υποβληθεί περίπου 33 τροπολογίες και ανάμεσα από αυτές και εξαιτία αυτών μάλλον, ο κύριος Μπρέντα λέει ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να παραμείνουμε στο ουσιαστικό θέμα της έκθεσης, το οποίο είναι με ποιον τρόπο μπορεί να βελτιωθούν οι διαδικασίες ηλεκτρονικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Όπως έχουμε ήδη συζητήσει στο παρελθόν. Δεν θα είχε νόημα να μπούμε σε λεπτομέρειες ή να συνδέσουμε, να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε αυτή τη συζήτηση με μια προσπάθεια ερμηνεία τη δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανταυτού, θα πρέπει να σκεφτούμε πώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε τι δυνατότητε που μα δίνει η ηλεκτρονική δημοκρατία και η τεχνολογία. Ο κύριος Πρέντα επίση έχει υποβάλει ε, για θέματα όπως τα ανοιχτά δεδομένα, η ιδιωτερότητα του δικτύου, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι σκόπιμο να μπούμε σε τέτοια γενικότερα ζητήματα, όπως για παράδειγμα η αδετερότητα του δικτύου, θέματα στα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφραστεί. Ε, έχουμε ήδη αναφέρει την σημασία που έχει η δυνατότητα, η πρόσβαση στο διαδίκτυο να είναι ανοιχτή και χωρί διακρίσει. Αυτό είναι σημαντικό την ηλεκτρονική δημοκρατία, αλλά πέρα από μια τέτοια γενική διατύπωση, διατύπωση δεν θα είχε νόημα να μπούμε στι λεπτομέρειε, στι τεχνικέ. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο το μήνυμά μα ότι αναφερόμαστε κυρίω στην ηλεκτρονική δημοκρατία. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει συνοχή με προηγούμενες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίω ε, αυτές που αφορούν στην αναθεώρηση του ε, εκλογικής νομοθεσίας για το Ευρωκοινοβούλιο. Θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικής πληροφορίε, πάντοτε λαμβάνοντας μέτρα τα οποία θα, ε, για να προστατεύσουν την ε, διαφάνεια της διαδικασίας. Θα πρέπει να ζητηθεί λοιπόν από τα κράτη-μέλη να διασφαλίζουν όταν χρησιμοποιούν τέτοιες δυνατότητες την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την μυστικότητα της ψηφοφορίας και την ασφάλεια. Βέβαια, ε, θα χρειαστεί καιρό μέχρι να έχουμε όλα τα δεδομένα στη διάθεσή μα, όλε τι ασφαλιστικέ δικλείδε, για να μπορούμε να πάμε προ μια κατάσταση που θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά η ψηφοφορία. οι συγκεκριμένες αρχές που θα πρέπει να ε, διασφαλίζονται αναφέρονται ε, συγκεκριμένα στην τροπολογία 19. Αναμένουμε μέχρι το τέλος του 2017 μία ε, πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και επίσης αναμένονται και μελέτες όμως πριν να προχωρήσουμε θα πρέπει να ε, γνωρίζουμε ποια είναι η άποψη των πολιτών, πώς ε, ε, αισθάνονται οι πολίτες απέναντι στην πιθανότητα να γίνονται ψηφοφορίες ηλεκτρονικά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα τροπολογία έχει υποβληθεί από τον ίδιο τον εισηγητή για την, την ηλεκτρονική ιδιότητα του πολίτη, την ηλεκτρονική συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, η citizenship. Ε, ο Πρέτα επίσης θεωρεί την πρόταση Ιταλών συναδέλφων να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή χάρτα για τα δικαιώματα στο ίντερνετ ως ενδιαφέρουσα θα, είχε, ε, θα ήταν σκόπιμο να προσπαθήσει να συμμετάσχει η Επιτροπή μας σε μια τέτοια διαδικασία όμως πρέπει να είμαστε ταυτόχρονα ρεαλιστές και να αναγνωρίσουμε ότι θα υπάρξουν προβλήματα σε μια τέτοια προσπάθεια γιατί συνδέεται με πολλές πτυχές της ευρωπαϊκής πολιτικής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν νομίζω ότι έχουμε άλλους ομιλητές. Θέλετε να μιλήσετε εσείς ε, εκ μέρους των Πρασίνων. Παρακαλώ. Μαξ, παρακαλώ. Ο σκιώδης εισηγητής των Πρασίνων, Μαξ Άντερσον, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να επισημάνω κάποια από τα βασικά στοιχεία στα οποία έχουμε υποβάλει τροπολογίες. Καταρχάς, δεν υπάρχει τρόπος να έχουμε πρόταση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ε, μέχρι το 2017 σε όλες ε, τις για ε, εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη μέχρι το 2019. Αυτό είναι αδύνατον. Γι' αυτό έχω υποβάλει τροπολογία για να τροποποιήσουμε την πρόταση αυτή. Όσον αφορά την ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία, υπάρχουν δύο διαφορετικές ε, γραμμές. Ε, υπάρχουν αυτοί που βλέπουν τα πιθανά πλεονεκτήματα και αυτοί που βλέπουν τα πιθανά προβλήματα. Θα πρέπει αυτά να τα ζυγίσουμε και ακολουθώντας μια προσεκτική προσέγγιση, θα έλεγα ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος ε, κυβερνοεπίθεσης, ειδικά στο παρόν περιβάλλον ασφαλείας, όπου κράτη-μέλη με οι υψηλέ ε, τεχνολογικέ δυνατότητε φαίνεται να θέλουν να παρέμβουν στα εσωτερικά άλλων χωρών. Υπάρχει λοιπόν τέτοιος κίνδυνο που συνδέεται με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίε. Χρειαζόμαστε ένα, ασφαλιστικό, ένα ασφαλές σύστημα και δεν ε, είναι κανένα σύστημα απολύτως ασφαλές. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι δηλαδή ότι τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ε, είναι περισσότερα από τους κινδύνους. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, να έχουμε προσεκτική προσέγγιση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτή την προσεκτική προσέγγιση στην έκθεση αυτή. Επίσης έχουμε κάποιες άλλες παρατηρήσεις, ε, για παράδειγμα την τροπολογία υπαριθμών 150. Προσπάθησα να διαβάσω όλες τις ε, τροπολογίες και όταν διάβασα το κείμενο σκέφτηκα πάρα πολύ καλή τροπολογία και μετά θυμήθηκα ότι εγώ την είχα συντάξει. Πάντα είναι ευχάριστο αυτό όταν συμβαίνει έχει να κάνει με την χρήση λογισμικού ανοιχτή πηγή και ανοιχτών προτύπων ε, στην ε, δημόσια διοίκηση. Και αυτό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση αυτή, γιατί αν θέλουμε μια ηλεκτρονική δημοκρατία που να λειτουργεί καλά, θα πρέπει να έχουμε συστήματα υπολογιστών ε, για την επικοινωνία με τους πολίτες. Θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να επιτρέπει στους πολίτες να χρησιμοποιούν έναν απλό υπολογιστή για να επικοινωνούν με την κυβέρνηση. Και όταν η κυβέρνηση δημοσιεύει πληροφορίες στο διαδίκτυο, οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν ε, να, το, να διαβάσουν τις πληροφορίες αυτές και γι' αυτό χρειαζόμαστε ανοιχτά πρότυπα. Τα ανοιχτά πρότυπα είναι θέμα δικαιοσύνης, ε, δημοκρατίας. Και επίσης ε, καλής πρακτικής αρχαιοθέτησης. Θα πρέπει να είναι δυνατό να διαβάσει κανείς τα έγγραφα του παρελθόντος. Δεν μπορούμε να έχουμε την κατάσταση όπου κάθε φορά που υπάρχει νέα εκδοχή του λογισμικού να μην μπορούμε πια να διαβάσουμε τα έγγραφα του παρελθόντος. Γι' αυτό το θέμα των ανοιχτών προτύπων είναι θέμα δημοκρατίας. Και το λογισμικό ανοιχτής πηγής θα πρέπει να χρησιμοποιείται ε, μερικές φορές έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Είναι πιο οικονομικό το λογισμικό ανοιχτή πηγής. Ε, και είναι πλεονέκτημα ότι απαιτεί και ανοιχτά πρότυπα. Αυτές είναι οι δύο κύριες τροπολογίες μου. Έχουμε υποβάλει και ένα σωρό άλλες πρακτικού τύπου τροπολογίες που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο των ε, ομάδων συμφερόντων, των λόμπις, ε, κάτι που ε, πάντα λέμε εμείς οι πράσινοι και διάφορες άλλες τέτοιες τροπολογίες. Μπορείτε να τις διαβάσετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Στο μεταξύ δεν ήρθε κανείς άλλος, δεν έχει ζητήσει κανείς άλλος το λόγο. Ραμόν, σου ξαναδίνω το λόγο, παρακαλώ. Bueno, Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα. Έχω σημειώσει πέντε, έξι ε, μεγάλες ενότητες ε, θεμάτων ε, στα οποία πρέπει να επικεντρώσουμε τη συζήτηση με τους κοιόδης συντάκτες και αυτό θέλω να κάνω στην επόμενη συνεδρίαση. Θέλω να δω λίγο το χρονοδιάγραμμα, να συνεδριάσω με όλους τους κοιόδης ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα έγγραφο ε, στο οποίο κατ' ουσίαν να υπάρχει συνένωση. Ε, σημειώνω καταρχάς, ε, George, κύριε Σέπφλιν, τις τροπολογίες που υπέβαλε το ΕΛΚ μέσω των κύριων Πρέτα και Μακάλιστερ. Γενικά να πω ότι θεωρώ ότι είναι λογικές. Ο κύριος Πρέγκα ναι, ανέκαθεν επέμεινε ότι πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα όταν κάνουμε τη διάγνωση της δημοκρατικής κρίσης. Ε, είναι σημαντικό αυτό προκειμένου ε, να μην ε, περιορίσουμε πάρα πολύ την αξιοπιστία του ίδιου του συστήματος. Εγώ είμαι ε, υπέρ ε, των ιδεών που μου έθεσε ο κύριος Πρέντα μέσω των τροπολογιών τους και θα τα συμπεριλάβω. Και ε, υπάρχει επίσης και σχέση με τη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε. Εδώ θα υπάρχει ένα σημείο τριβής με τροπολογίες που υπέβαλαν κάποιες πολιτικές ομάδες, κυρίως ο κύριος Καστάλτο και η κυρία Αντινόλφη, όσον αφορά την αμεσοδημοκρατία διότι υπάρχει πάντα δυνατότητα ε, να ζητήσουν κάποιες ομάδες, κυρίως ε, τώρα τελευταία, να επιτύχουμε βελτίωση της δημοκρατίας μέσω δημοψηφισμάτων, μέσω άμεσης διαβούλευσης με τους πολίτες. Αυτό το οποίο θα αποκαλούσαμε άμεση δημοκρατία. Κάτι που κατά την άποψή μου δεν μπορεί να αποτελεί εναλλακτικό σύστημα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Εγώ πιστεύω ότι η εμπειρία των τελευταίων ετών ε, καταδεικνύει ότι η λεγόμενη άμεση δημοκρατία δεν είναι ένα πιο αγνό και τελειότερο σύστημα από την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Εγώ αντιθέτως φρονώ ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι πολύ πιο αχνό σύστημα από την άμεση δημοκρατία. Αυτό δεν αποκλεί το ενδεχόμενο πότε πότε να μπορούμε να προσφύγουμε σε συστήματα δημοψηφίσματος κλπ. Αλλά επαναλαμβάνω η εμπειρία αποδεικνύει ότι τα δημοψηφίσματα εν γέννη συσσωρεύουν ε, απλές απαντήσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα. Και δεν είναι αυτός πάντα ο καλύτερος τρόπος ε, να ακούσουμε τη γνώμη των πολιτών. Ε, όπως και να έχει τέλος πάντων, εδώ κάνουμε μια συζήτηση. Εγώ τίνω μάλλον προς τη μεγαλύτερη σοφροσύνη για τη συζήτηση αυτή. Και υπάρχει ένα θέμα το οποίο μόλις έθεσε ο κύριος Άντερσον και είναι πολύ σημαντικό και εμείς θα το συμπεριλάβουμε όσον αφορά τον ανοιχτό κώδικα ή αυτό το οποίο ε, αποκαλούμε ελεύθερο λογισμικό, δηλαδή οι πολίτες να μην εξαρτώνται από συγκεκριμένη τεχνολογία λογισμικού, ώστε η πρόσβαση τους ε, στις διάφορες μορφές τεχνολογίας να είναι απόλυτα ελεύθερη. Ε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν υπήρχε στην έκθεση, θα το συμπεριλάβουμε. Υπάρχουν αρκετέ τροπολογίες ε, και θα ήθελα να το προτείνω στον κύριο Σέπφλιν όσον αφορά ε, τι πρωτοβουλίε των πολιτών. Την ε, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, στην οποία επαναλαμβάνονται όλα τα πράγματα τα οποία έχουμε πει για τις δυνατότητες βελτίωσης του συστήματος της πρωτοβουλίας των πολιτών. Θεωρώ όμως ότι αυτό είναι εκτός τόπου και χρόνου, γιατί τα έχουμε πει αυτά ε, στις εκθέσεις ε, που εκπονήθηκαν ε, από τον ίδιο τον κύριο Σόπφλιν και ενέκρινε η Επιτροπή μας όσον αφορά τον τρόπο να βελτιωθεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση νομίζω για το κατά πόσον θα πρέπει να ζητήσουμε ε, ρύθμιση του διαδικτύου ή όχι. Και εδώ νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση ουσία. Υπάρχουν αρκετέ τροπολογίε, οι οποίες επιμένουν ότι το δίκτυο πρέπει να τύχει ρύθμιση. Και αυτή είναι μια συζήτηση που θεωρώ ότι δεν είναι αφηρημένη συζήτηση. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μας υποχρεώνει να σκεφτούμε και λίγο κατά πόσον είναι δυνατόν κάτι τέτοιο και αν συστήνεται κάτι τέτοιο από πολιτική σκοπιά. Ε, υπάρχουν αρκετές ε, προτάσεις η έκθεση να συμπεριλάβει και την ε, διαφορά που υπάρχει μεταξύ της τεχνολογίας της πληροφορίας ε, και των ατομικών δικαιωμάτων. Ε, την τιμή, ε, η κυρία Μπρέσο για παράδειγμα έχει κάποιες πρωτοβουλίες που ζητούν η χρήση των τεχνολογιών να συνοδεύεται και από συστήματα προστασίας των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Ε, το δικαίωμα στη για να δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο γνωρίζετε όλοι, και βεβαίως και η ε, προστασία του καθενός από ένα δίκτυο, το οποίο γνωρίζουμε όλοι ότι γεννά μια πολύ σοβαρή ρήξη ε, για αυτό το οποίο αποκαλείται τώρα ε, ε στα αλήθεια, δηλαδή διάφορα πράγματα τα οποία τείνουν να πιστεύονται ως αληθή λόγω της μαζικής χρήσης του διαδικτύου. Και όταν αυτό επηρεάζει τη ζωή των ατόμων ε, και τα δικαιώματά τους, θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματά τους. Αυτό θα πρέπει να το περιλάβουμε στην έκθεση. Υπάρχουν αρκετές... τροπολογίες που ζητούν να δούμε τους κινδύνους του μονοπωλίου της κοινή γνώμης όταν ασκείται μέσω του διαδικτύου από τομεακά λόμπι, από οργανώσεις οι οποίες αναλαμβάνουν ε, να εκπροσωπήσουν αυτό το οποίο φαίνεται ότι είναι η μαζική άποψη των πολιτών. Αυτό το βλέπουμε όλοι, γιατί να σας τα πω εγώ, όλοι κάθε μέρα λαμβάνουμε χιλιάδες ε, θέσεις και απόψεις οι οποίες εκπροσωπούν τους πολίτες, μεν, αλλά ε, μπορεί να τις χειραγωγεί απλώς ένα μηχάνημα που απλώς μας διαβάζει ονόματα ανθρώπων που είναι υπέρ της τάδε θέσης ή που συστήνουν να ψηφίσουμε το τάδε ή το δίνα. Δεν μπορούμε να μην το επισημάνουμε εδώ στην έκθεση. Το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχει ο κίνδυνος συγκεκριμένες οργανώσεις που χειραγωγούν τις διάφορες μορφές επικοινωνίας να μας διαβιβάσουν μια άποψη η οποία αντικειμενικά δεν θα είναι η άποψη των πολιτών αλλά θα είναι απλώς η ε, τεχνική συσσόρευση των απόψεων κάποιων πολιτών. Και επίσης υπάρχει και κάτι το οποίο ε, σχολίασε και ο κύριος ε, Σόπφλιν όσον αφορά το δικαίωμα αναγνώριση της πρόσβασης στο διαδίκτυο ως θεμελιώδης δικαίωμα. Οι Ιταλοί κινήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση, εγκρίθηκε και από το κοινοβούλιο τους ε, μία μορφή χάρτας των δικαιωμάτων πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ειλικρινά πιστεύω ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε αυτή την ιδέα ότι αυτό στο μέλλον, εάν δεν είναι ήδη, θα γίνει θεμελιώδης δικαίωμα. Ε, Βεβαίω, ε, η συγκεκριμένη γνωμοδότηση προτείνει απλώς ιδέες και ε, προσανατολισμούς. Επομένως, ίσως πρέπει να συμπεριλάβουμε και αυτή την άποψη. Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι όπως σα υπενθύμησα, η πρόθεσή μου είναι να συνεδριάσω με του ισχυωδείς συζήτητες. Καταρχάς, θα του στείλω τι συμβιβαστικέ προτάσεις ε, στις οποίες νομίζω ότι αντανακλώνται οι θέσει τους, ώστε να μπορέσουν <coughs> να συμφωνήσουν, αν θέλετε, με τη νέα διατύπωση ε, και αυτή τη στιγμή ε, μπορέσουμε να συνεργαστούμε ως προς το σχέδιο κειμένου που θα του στείλω. Θα οργανώσω μια συνεδρίαση και επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε να προτείνω τον Ιανουάριο να ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση διότι νομίζω ότι ε, είναι ενδιαφέρουσα για το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Χαμόν. Να σας ενημερώσω ότι η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για την συνεδρία σήμα στις 30 και 31 Ιανουαρίου. Και πράγματι, όπως είπαστε, εν τω μεταξύ, από τώρα μέχρι τις 30-31 Ιανουαρίου θα οργανώσετε τις συναντήσεις με τους Χιώδης, με τη βοήθεια της Γραμματείας έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για την ψηφοφορία τον Ιανουάριο. Και πράγματι ελπίζω όπως και εσείς ότι αυτή η έκθεση θα είναι ενδιαφέρουσα και ουσιαστική. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσια διάταξης, το πέμπτο, για την γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνδευματικών Εγωθέσεων για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων. Ε, είμαι ίδια η συγγήτρια και επίσης, από ό,τι φαίνεται, μόνο η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων θα υποβάλει νομοδότηση. Αυτό, αυτή η πρόταση είναι ο τρίτος πυλώνας για την ολοκλήρωση της ε, Τραπεζικής Ένωσης, η οποία, όπως γνωρίζετε, προσπαθεί να προλάβει την ε, κατάσταση κατά την οποία οι πολίτες θα έπρεπε να αναλάβουν να πληρώσουν για τα προβλήματα, για τα λάθη, ε, για τι λανθασμένε επιλογές τραπεζών. Η συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων στην ΕΚΟΝ ήταν δύσκολη, έχει παραμείνει στην ημερήσια διάταξη για πολύ καιρό ε, συζητηθεί ε, και καθυστερήσει πολλές φορές και είναι πιθανό να, υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση. Ο προγραμματισμός αυτή τη στιγμή της ΕΚΟΝ είναι να ε, συζητηθεί τέλος Ιανουαρίου. Ε, η διαδικασία που γνωρίζετε είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποβάλει την γνωμοδότησή κάνει μάλλον τις παρατηρήσεις του πάνω στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα επίσης να σας ε, φυστήσουν στην προσοχή στο γεγονό ότι οι τροπολογίες από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων πρέπει να περιοριστούν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Ε, άλλα θέματα ε, θα πρέπει να συζητώνται ή να υποβάλλονται στην κατ' ουσίαν αρμόδια Επιτροπή. Εδώ την οίκον δηλαδή. Επομένως, εγώ θα στεκόμουν σε τρεις σημαντικές αρχές που αφορούν την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, τις οποίες η αρμοδιότητα είναι η συνταγματική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο είναι η ασφάλεια δικαίου, το δεύτερο είναι η ισότητα των κρατών μελών. Ε, όσον αφορά την ασφάλεια δικαίου, θα πρότεινα να υπάρξει μια συγκεκριμένη αναφορά στο τι συμβαίνει όταν ένα ε, εθνικό σύστημα εγγύησης καταθέσεων το οποίο συμμετέχει στο ευρωπαϊκό αποτυγχάνει ή μάλλον δεν, δεν ε, πληρεί τις προϋποθέσεις του ευρωπαϊκού συστήματος. Η διαδικασία την οποία προτείνει η Επιτροπή σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να αποκλείεται ε, το εθνικό εκείνο σύστημα από το, την, την κάλυψή του από τον μηχανισμό έντις. Κατά την άποψή μου αυτό δεν είναι σωστό από την άποψη της αρχής της αναλογικότητας. Εμείς θα θέλαμε το σύστημα το οποίο θα δημιουργηθεί ε, να εξασφαλίζει την ασφάλεια δικαίου, να είναι προβλέψιμο και αυτό σημαίνει να υπάρχει μια κάποια διαδικασία πριν φτάσουμε στις κυρώσεις. Πριν φτάσουμε στην ε, στον αποκλεισμό του εθνικού συστήματος από το ευρωπαϊκό, από το ΕΔΙΣ. Για παράδειγμα, σε πρώτο στάδιο να προβλέπετε κάποιο πρόστιμο. Και για να υλοποιηθεί αυτό στην πράξη, προτείνω με μια τροπολογία μου να δοθεί δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω μια πράξη εξουσιοδότηση να δημιουργήσει ένα τέτοιο σύστημα ε, κυρώσεων. Δεύτερο θέμα το οποίο θα ήθελα να αναδείξω είναι τι θα συμβεί στην περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος το οποίο δεν έχει ο νόμισμά του το ευρώ συμμετάσχει στο σύστημα, ενταχθεί στο σύστημα. Στην αρχική πρόταση της Επιτροπής προβλέπεται μια διαδικασία ε, με την οποία μπορεί να ε, ε, μεταφερθούν κονδύλια προς το εθνικό σύστημα εγγύησης καταθέσεων εάν μια χώρα φύγει από την, από την Τραπεζική Ένωση. Προβλέπετε λοιπόν τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση, αλλά δεν προβλέπετε πώ το κράτο μέλος θα ενταχθεί στο έντι και στο σύστημα εγγύηση. Αυτό λοιπόν που προτείνω με την, στην, στην εισήγησή μου είναι να υπάρχει ένα σύστημα και για την είσοδο και για την έξοδο. Phase in και phase out. Επίσης όσον αφορά την λογοδοσία. Προτείνω να καταγραφεί με σαφήνεια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποχρεούται να ενημερώνει και να διαβουλεύεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οποτεδήποτε ε, γίνεται κάποια μεταβολή στο, ε, στο, στο, στο έντις, στο στους πόρους που είναι διαθέσιμοι για το ΕΝΤΙΣ. Αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται κάποια συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε αποκλειστεί και πιστεύω ότι είναι λάθος και θα πρέπει να αλλάξει. έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ε, σύνδεση Μάλλον, ακόμα μια πρόταση αφορά στον τρόπο με τον οποίο τα, οι αρχές που θα διαχειρίζονται το έντις θα συνεργάζονται με τις αρχέ ε, τι εθνικέ. εποπτικές. Πιστεύω ότι σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να συμμετέχουν λοιπόν και οι διαχειριστές του έντις. Και επίσης να δοθεί η δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όχι μόνο στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συγκαλεί έκτακτη ε, συνάντηση, συνέλευση του ΕΔΙΣ. Αυτή τη στιγμή αυτό το δικαίωμα προβλέπεται μόνο στην Επιτροπή, ενώ εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να το έχει και η ΕΚΤ. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι στις 7 Δεκεμβρίου 6 το απόγευμα. Και η ψηφοφορία προτείνουμε να γίνει στις 30 Ιανουαρίου. Αυτή η πρόταση για αυτές τις προθεσμίες γίνεται επί τη βάση της διαδικασίας που προβλέπει να ακολουθήσει και η εικόνα. Τώρα έχουμε το πρόβλημα. Μόνο η Mercedes είναι παρούσα και θα ήθελε να λάβει το λόγο για το θέμα αυτό ενώ έχει ήδη προσέλθει ο πρέσβης ε, Γιώφτσικ, όπως σας είχα ενημερώσει, ο κύριος Γιώφτσικ θα πρέπει να φύγει στις 10. Γι' αυτό θα πρότεινα το εξή, μια και ορισμένα μέλη Εθνικών Κοινοβουλίων έχουν ήδη προσέλθει και καλώς ορίσατε. Αναρωτιέμαι τι να κάνω, να ξεκινήσω τώρα την συνάντηση επισήμως όχι. Απλώς, ε, κύριε Πρέσβη, δεν ήθελα να καταχρωστώ το χρόνο σας, επομένως θα δώσω το λόγο στο πρέσβη. Ευχαριστώ. Όταν μπορείτε. Σας ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη ε, για την τροποποίηση αυτή της ημερήσιας διάταξης. Καταλαβαίνετε όμως πλησιάζει το τέλος της Προεδρίας μας και θα πρέπει σε λίγο να σας εγκαταλείψω για να ε, παρευρεθώ στον τριμερή διάλογο στις 10 η ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Ε, είναι ε, πολύ ευχαριστή ευκαιρία για μένα να μπορέσω να σας ε, μιλήσω εκ μέρους ε, της Σλοβακικής Προεδρίας στην συνάντηση αυτή ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα ήθελα να σας πω πόσο η Προεδρία μας εκτιμά τη συνεργασία μαζί σας και προσωπικά με σας και με τα μέλη της Επιτροπής σας. Η συνεργασία μας είναι πολύ καλή, πολύ επικοδομητική. Και ήδη είχα παρευρεθεί εδώ στη συνεδρίασή σας ε, τον ε, Σεπτέμβριο, αλλά σας συνάντησα και σε ταξίδι στην Βρατισλάβα αρχές Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Να πω λίγα λόγια για την Προεδρία μας γενικά. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Απομένει ακόμα δουλειά να γίνει τις ε, τελευταίες εβδομάδες. Προσπαθούμε λοιπόν ε, να εργαστούμε σκληρά για να ε, πραγματοποιήσουμε τις φιλοτοξίες μας, όπως σας είπα στην αρχή. Να σας πω κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τη γενικότερη εικόνα. Η διάσκεψη κορυφή της Πρατισλάβα πραγματοποιήθηκε μέσα Σεπτεμβρίου, ουσιαστικά όρισε την Προεδρία μας. Το βασικό μήνυμα ήταν πώς να επανέλθει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον δρόμο της μετά από το δημοψήφισμα του Brexit. Υπάρχει λοιπόν ο δικός χάρτης της Πρατισλάβα, ο οποίος επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους στόχους από αποτελέσματα πράγματα που έχουν σημασία για τους πολίτες μας. Ε, και η Προεδρία μας διαμορφώθηκε με επίκεντρο αυτό. Ελπίζουμε λοιπόν ε, τον Δεκέμβριο να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, επικεντρωνόμαστε στην εφαρμογή ε, της ε, Ευρωπαϊκής ε, Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, μιας πρότασης που υιοθετήθηκε στο Συμβούλιο και τώρα έχει έρθει η ώρα εφαρμογής της πρότασης αυτής. Ελπίζουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς να μπορούμε να δείξουμε ότι δεν είναι κάτι που παραμένει αποκλειστικά στο χαρτί. Ελπίζουμε μέσα σε αυτό το εξάμεινο να προχωρήσουμε όσον αφορά την επικύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα από τα συμβαλώμενα μέρη Και ε, έχουμε και την συνάντηση των μερών ε, στο Μαρακές. Ε, δεν θέλω να αναφερθώ πολύ στην ΣΥΤΑ. Ήταν δύσκολες οι διαπραγματεύσεις. Καταφέραμε όμως να ολοκληρώσουμε την διαδικασία της υπογραφής. τώρα βρίσκεται ακόμα στο Κοινοβούλιο η πρόταση αυτή. Είναι όμως πολύ σημαντικό βήμα ε, όσον αφορά την εμπορική πολιτική μας. Επίσης ε, καταφέραμε να συμφωνήσουμε όσον αφορά τον αποκλεισμό στο Συμβούλιο. Ε, πρόκειται λοιπόν για κομμάτια του πάζελ. και με την κυρία Γεωργίευα είχαμε καλή συζήτηση για τον προϋπολογισμό και την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Όσον αφορά λοιπόν ε, το θεματολόγιο της ε, Επιτροπής ΑΦΚΟ, έχουμε και εδώ κάποια σημαντικά αποτελέσματα. Προχωρήσαμε όσον αφορά τον, τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου. Θα μπω σε λεπτομέρειε αργότερα. Συμφωνήσαμε με το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά ε, το δικαίωμα εξέταση των πραγμάτων του Κοινοβουλίου και επίση ετοιμάζουμε την ε, διαθεσμική συμφωνία ε, σχετικά με το Μητρό Διαφάνειας. Είχαμε λοιπόν κάποιες χρήσιμες συναντήσεις ε, και για τα θέματα αυτά. Πιο αναλυτικά όσον αφορά το εκλογικό νόμο. Το Συμβούλιο συμμερίζεται τον στόχο του Κοινοβουλίου ε, να αυξήσει το ενδιαφέρον και την ε, συμμετοχή στις εκλογές, ε, στις ευρωεκλογές. Και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την πρόταση, προσπαθούμε να χαρτογραφήσουμε την κατάσταση και την πρόταση του Κοινοβουλίου. θα είναι δύσκολο να πετύχουμε συμφωνία, ομοφωνία ανάμεσα στα κράτη-μέλη όσον αφορά κάποια στοιχεία της ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να είμαι απόλυτα ειλικρινή. Προσπαθήσαμε όμω ε, να εντοπίσουμε ε, κάποια στοιχεία τα οποία να μπορούν να αποτελέσουν βάση για πρόοδο και να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο πλαίσιο για την διεξαγωγή των ευρωεκλογών. Ω Προεδρία, ο ρόλο μα είναι να διευκολύνουμε τη συζήτηση εντό του Συμβουλίου και να πετύχουμε συνένεση πάνω στα στοιχεία αυτά και πάνω σε κάποια σημεία τη πρόταση. Είχαμε εντατικέ συζητήσει σε επίπεδο ομάδα εργασία. Θα συζητήσουμε μάλιστα το θέμα αυτό αύριο στην Κορεπέρ. Θα συζητήσουν οι πρέσβεις δηλαδή και ελπίζω μετά να μπορέσω να επιστρέψω εδώ στην Επιτροπή σας και να σας αναφέρω ποια είναι τα πιθανά στοιχεία για μια μελλοντική συμφωνία. Ξέρω ότι ο χρόνος τρέχει. Γι' αυτό η Προεδρία μας ε, ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα αυτό και ελπίζουμε να έχουμε αποτελέσματα μέσα στο πρώτο εξάμεινο της επόμενης χρονιάς, να έχουν ολοκληρωθεί δηλαδή οι συζητήσεις. να πω όμως εδώ ότι ο στόχος είναι να αυξήσουμε τη συμμετοχή ε, των ε, ψηφοφόρων στις εκλογές. Να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες, ένα καλύτερο πλαίσιο. Σημαντικό είναι όμως ότι οι ευρωεκλογές ε, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατικής διαδικασίας εντός των κρατών μελών. Πιστεύουμε ότι με κάποιες νομοθετικές προσαρμογές θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό, αλλά βέβαια ε, είναι πολύ σημαντική η ε, συμμετοχή των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων. Όσον αφορά το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαίρομαι που συμφωνούμε με το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω στο θέμα αυτό. Είχαμε συνάντηση όπου συμφωνήσαμε για να ξεκινήσουν οι επίσημες διαπραγματεύσεις είναι απαραίτητο να παρουσιαστεί η συγκεκριμένη διατύπωση από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναγνωρίσαμε επίση ότι η διαδικασία ε, σύνταξη του κειμένου αποτελεί αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου. Συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε στην ε, επίσημη ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στις ε, νομικές υπηρεσίες το ε, Συμβούλιο, το, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο και στόχος μας είναι να εντοπίσουμε εδώ τα ε, νομικά και θεσμικά θέματα. Υπάρχει όμως κοινή κατανόηση. Θέλουμε λοιπόν να διευκολύνουμε τις επαφές ανάμεσα στις νομικές υπηρεσίες, κάτι που μπορεί ε, να ξεκαθαρίσει και το πλαίσιο εντός του οποίου μπορούμε να προχωρήσουμε. Να καλέσω λοιπόν και εσά ε, να οργανωθεί όσο γίνεται πιο σύντομα αυτή η συνάντηση των ε, νομικών υπηρεσιών ε, όσον αφορά την μελλοντική ανάπτυξη της Ένωση. Και αναφέρομαι στην έκθεση του κυρίου Μπροκ και της κυρίας Μπρέσο σχετικά με την βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι και στην έκθεση του κυρίου Φερχόφστατ για τις ε, προσαρμογές ε, στην παρούσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιβεβαιώνω ότι εμείς ως ε, Προεδρία προσβλέπουμε να λάβουμε τις εκθέσεις αυτές μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσα στο πρώτο εξάμεινο της επόμενης χρονιάς δηλαδή. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκλησή σας και προσπάθησα να σας δώσω μια εικόνα σχετικά με το πού βρισκόμαστε ως Προεδρία. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριο Πρέβρη, Πρέσβη για τους συναδέλφους που μόλις ήρθαν. Επειδή ο πρέσβης Πίτερ Γιάκη, ο κοφτής της Σλοβακικής Προεδρίας, έχει κάποιες υποχρεώσεις ε, για τριμερή διάλογο. Ε, χρειάστηκε να ακούσουμε την άποψή του και τόσο έχει να μας πει πριν από τη συνεδρίαση. Για όσους από εσά λοιπόν ήρθαν λίγο αργότερα, ακούσατε κάποιο τμήμα, αλλά δεν ε, είχαμε άλλο τρόπο να ακούσουμε τα της Προεδρίας από τον Πρέσβη. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέσβη λοιπόν και ελπίζουμε ότι όλα εκείνα που μας αναφέρετε θα μπορέσουμε να τα ολοκληρώσουμε. Ε, μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι για πολλά πράγματα δεν έχουμε ολοκληρώσει ε, στη διάρκεια της Προεδρίας σας και δεν θα ολοκληρωθούν στη διάρκεια της Προεδρίας σας, αλλά είχαμε και τη δυνατότητα μαζί σας όσον αφορά τον εκλογικό νόμο να συζητήσουμε και το δικαίωμα στην έρευνα. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που ήσασταν ε, μαζί μας και μας στηρίξατε σε αυτά τα δύσκολα θέματα. Σας ευχόμαστε λοιπόν ό,τι καλύτερο για τους τελευταίους ε, εβδομάδες της Προεδρίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε επισήμως ε, τώρα τη συνεδρίασή μας. Θα ήθελα καταρχάς να αποχαιρετήσω τον ε, πρέσβη Γιάβορτσι και ε, να καλωσορίσω ε, τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Αντιπρόεδρο, την κυρία Κλεισταρίνα Γεωργίευα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι δυστυχώς υπάρχει μία ψηφοφορία στο Σλοβακικό Εθνικό Συμβούλιο. επομένω ο συνάδελφο, ο πρόεδρο ε, της Επιτροπής ε, Συνταγματικών Υποθέσεων, ο κύριος Ρόμπερτ Μάντε, ο οποίο υποτίθεται ότι θα συμπροεδρεύει μαζί μου σήμερα, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Επίση, οι συνάδελφοι από την ε, Πορτογαλική Εθνοσυνέλευση έχουν κάτι αντίστοιχο, ψηφοφορία για τον προπολογισμό του 2017 σήμερα και μας ζήτησαν να σας εξηγήσουμε γιατί δεν μπορούν να παρευρεθούν. Θα ήθελα επίσης να πω δύο λόγια και να σας υπενθυμίσω ε, γιατί είμαστε εδώ. Διότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκμεταλλευόμαστε όλες τις πιθανές ε, πλατφόρμες ε, που έχουμε ε, συστήσει ή θα μπορούσαμε να συστήσουμε προκειμένου να γίνει ένας πολιτικός διάλογος με τα Εθνικά Κοινοβούλια και η ΑΦΚΟ έχει οργανώσει κάθε χρόνο, οργανώνει μάλλον αυτή τη συνεδρίαση με τη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια για να συζητήσει θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για το πολιτικό θεματολόγιο της Επιτροπής Δαγματικών Υποθέσεων. Θεωρούμε ότι μέσω αυτού του δικτύου των εθνικών βουλευτών και των ευρωβουλευτών μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες, μπορούμε να συνεισφέρουμε στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών καλύτερα και επίσης ε, μπορούμε να έχουμε και μεγαλύτερη επιρροή στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών ε, σε εθνικό επίπεδο. Επομένως ελπίζω ότι η σημερινή συνεδρίαση θα αποτελέσει μια ακόμα ευκαιρία ε, σε αυτή την προσπάθεια να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων ε, των πολιτών ε, στα διάφορα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω και να σας ανακοινώσω στην ουσία ότι κατά πάσα πιθανότητα θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας το πρώτο εξάμεινο του 2017 γιατί ο συνάδελφος ο Πάολο Ρανζέλ αυτή τη στιγμή ασχολείται με μια έκθεση εφαρμογής, όπως αποκαλείται, ε, που στόχο έχει να εξετάσει την εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης όσον αφορά το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα μπορέσει να σας επισκεφθεί όλους, αλλά ίσως θα ήταν και πιο ε, χρήσιμο να σας καλέσουμε εδώ και να γίνει και μια διακοινοβουλευτική συνεδρίαση για το θέμα αυτό στο πρώτο εξάμεινο του 2017. Ώστε να μπορέσουμε λοιπόν να σας ρωτήσουμε με ποιο τρόπο θα θέλατε να γίνει η συμμετοχή σας στη συζήτηση για τα θέματα αυτά, τα οποία είναι ε, τμήμα της έκθεσης. Η σημερινή συνεδρίαση, όπως γνωρίζετε, το εξή. Το πρωί θα γίνει συζήτηση για δύο εκθέσεις, οι οποίες αναφέρθηκαν από τον πρέσβη Γιάβορτσικ και είναι τμήμα της συνεργασίας μεταξύ ε, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Η μία αφορά τον κανονισμό για το δικαίωμα ε, έρευνας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Και ε, ε, το άλλο είναι ο εκλογικός νόμος ε, του 1976. Στόχος αυτών των δύο προτάσεων είναι να να μπορέσουμε να συμμετέχουμε, να επηρεάσουμε και να δούμε και θέματα τα οποία είναι εγκάρσια το δικαίωμα της εξέτασης που είναι κάτι το οποίο απαιτεί συνεργασία αλλά φυσικά και ο εκλογικός νόμος ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός στα πλαίσια του δημοκρατικού ελλείμματος όπως το αποκαλούμε. Θα θέλαμε να προβάλλονται περισσότερο οι εκλογές, να είναι πιο ευρωπαϊκές και να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή. Και το απόγευμα θα γίνει συζήτηση για τη μελλοντική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σχέση που υπάρχει με τις θεσμικές και συνταγματικές ε, πτυχές. Θα συζητήσουμε λοιπόν ε, θέματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε στο παρόνομικό πλαίσιο, επομένως μπορούμε να συζητήσουμε θέματα που αφορούν ε, την έκθεση του Έλμαρ Μπρόκ και της Mercedes Μπρέσο για το πώς μπορεί να προχωρήσει η Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα θα μένει και εντός του πλαισίου των υφιστάμενων συνθήκων και ε, το δεύτερο τμήμα της συζήτησης ε, θα είναι αφιερωμένο στην έκθεση του Γκίφερ Χόφστατ, η οποία εξετάζει παραπέρα από τον, ε, τις παρούσες συνθήκες και βλέπει τις θεσμικές και σταγματικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν προκειμένου η Ευρώπη να αποφέρει τους καρπούς που υποτίθεται ότι πρέπει να αποφέρει για τους πολίτες και φυσικά και τι αλλαγές θα χρειαστούν στις συνθήκες προκειμένου να επιτευχθεί αυτό. Οι εκθέσεις αυτές είναι τμήμα της ε, διαδικασίας ε, της διαμόρφωση της άποψη του Κοινοβουλίου για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο, ο χάρτης πορείας της Πλατισλάβα δηλαδή, στον οποίο αναφέρθηκε ο πρέσβης ε, το τι γίνεται επίσης ε, στο Συμβουλίο όσον αφορά τα πλαίσια της ε, επαιτίου της συνθήκης της Ρώμης που θα γιορταστεί το Μάρτιο και τις εκδηλώσεις που θα γίνουν το Μάρτιο στη Ρώμη και στα πλαίσια του τι περιμένει με ανυπομονησία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έλεγα, το ε, έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Λευκή Βέβλο, τα επόμενα βήματα λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μελλοντική βελτίωση της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς ε, πιστεύω ότι πρέπει να ακουστεί και η φωνή μας σε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα επίσης να σας αναφέρω και πώς θέλουμε να οργανώσουμε αυτές τις συζητήσεις. Υπάρχει ένα έντυπο μπροστά σας. Μπορείτε να το συμπληρώσετε για κάθε τμήμα της συνεδρίας και θα φροντίσουμε φυσικά να κατανέμουμε το χρόνο αγόρευσης ε, δίκαια και θα ήθελα να σας ζητήσω λοιπόν ανάλογα με το θέμα στο οποίο θα θέλετε να μιλήσετε, να συμπληρώσετε το έντυπο και να το δώσετε... Ε, κάποιος θα, το, θα γύρει στην αίθουσα και θα το ε, μαζέψει. Θα δούμε πόσο χρόνο έχουμε και πόσο χρόνο μπορούμε να σας αφιερώσουμε. Είσαστε εξοικειωμένοι άλλωστε με αυτόν τον τρόπο εργασίας, διότι αυτό κάνουμε και στην ΚΟΖΑ και σε άλλες συνεδριάσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτά λοιπόν είναι είδη και τώρα θα ήθελα να ε, ζητήσω από τα μέλη του Κοινοβουλίου ε, τους εθνικούς βουλευτές, ε, την κυρία Επίτροπο βεβαίως και τον Επίτροπο Γιάβρουτσικ αν δεν έχει άλλες υποχρεώσεις να γευματίσετε μαζί μας. Θα θέλαμε να έχουμε ένα κοινό γεύμα μετά από την πρωινή συνεδρία στο μηδέν του κτηρίου, στο Ισόγειο. Ε, στο ε, εστιατόριο των βουλευτών. Ε, αυτά λοιπόν εισαγωγικά και τώρα να δώσω το λόγο στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Χούμπνερ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να απευθυνθώ σε εσάς σήμερα το πρωί εκπροσωπώ και τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς, ο οποίος πολύ θα ήθελε να παρευρίσκεται, αλλά σήμερα οργανώνει τον, ε, τον διαθρησιακό διάλογο και ζήτησε να παρευρίσκεται εκ μέρους της Επιτροπής και ζήτησε από εμένα να εκπροσωπήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αξιότιμα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα ξεκινήσω με μία διαπίστωση που δεν θα σας εκπλήξει. Ο κόσμος μας αλλάζει και πολύ γρήγορα. Πολλές από τις αλλαγές είναι προς το καλύτερο. Είναι θετικές. Το ΑΕΠ το συνολικό που παράγεται παγκοσμίω σήμερα είναι 83 εκατομμύρια δολάρια. Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο που ευημερεί περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι την τελευταία, τις τελευταίες δύο δεκαετίες ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι έπαψαν να βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Η τεχνολογία έχει αλλάξει και συνεχίζει να αλλάζει συνεχώς την καθημερινότητά μας. κοιτώ την εγγονή μου και διαπιστώνω πόσο άλλαξαν τα πράγματα από τότε που εγώ ήμουν μικρή. Τη λέω όταν εγώ είχα την ηλικία σου, είναι πέντε χρονών, δεν είχαμε τηλεόραση, δεν υπήρχαν υπολογιστέ. Και με κοιτάει με απορία και μου λέει, α, δηλαδή δεν είχατε μόνο iPad, έτσι. αν σκεφτούμε πώς εμείς ήμασταν στο σχολείο και πώς σήμερα οι μαθητές μαθαίνουν, οι αλλαγές είναι τεράστιες. Ή επίσης ο τρόπος με τον οποίο ε, παρέχονται υπηρεσίες. Οι αλλαγές είναι δραματικές και γνωρίζουμε όμως ότι αυτές οι αλλαγές δεν είναι μόνο θετικές. Η διασύνδεση έχει η μεγαλύτερη ε, διασύνδεση έχει δώσει τη δυνατότητα σε εμπορεύματα, σε, ε, σε, στις, πληροφορίες να διαδίδονται, αλλά ανάμεσα σε αυτές τις πληροφορίες είναι και ε, ιδεολογίες που κηρύσουν ε, τη βία, για παράδειγμα. οι άνθρωποι επίση μετακινούνται πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν αλλαγές όλες αυτές έχουν οδηγήσει σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πολύ πιο ε, ευαίσθητος από ό,τι στο παρελθόν, εύθραυτος από ό,τι στο παρελθόν. Και το βλέπουμε αυτό ε, διαπιστώνοντας ε, τις συγκρούσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή και ένα ακόμα στοιχείο που έχει, που έχει αποκτήσει δυνατότητα να ε, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο είναι οι οικονομικές κρίσεις. Μια κρίση στην Ασία την επόμενη μέρα το πρωί θα γίνει αισθητή στην Ευρώπη. Είχαμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε πολλέ κρίσει. τελευταία 7 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έκανε τίποτε άλλο από το να αντιμετωπίζει τη μία κρίση μετά την άλλη. Η οικονομική κρίση, η κρίση τη Ευρωζώνη, η κρίση στην Ελλάδα, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, μετά το προσφυγικό. Και τώρα βρισκόμαστε ενώπιον πολιτικών ε, κρίσεων, όπω για παράδειγμα το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες αυτές οι διαπιστώσεις μας οδηγούν στο να αντιληφθούμε ότι υπάρχει ανάμεσα στους πολίτες μας μια ανησυχία την οποία έχουν εκμεταλλευτεί ορισμένοι για να την αξιοποιήσουν ε, προ όφελο του λαϊκισμού. Βεβαίω αυτή την ανησυχία θα πρέπει να τη λάβουμε σοβαρά. Οφείλουμε να τη λάβουμε σοβαρά. Όμω βλέπουμε την άνοδο του λαϊκισμού παντού. Και αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη η πλειονότητα των πολιτών πιστεύει ότι οι καλές εποχές πέρασαν και ότι αυτό που ανοίγεται μπροστά μας είναι μια εποχή αβεβαιότητας. Και αυτή η κατάσταση μας οδηγεί πολύ συχνά να ξεχνούμε τα θετικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως, για παράδειγμα, το γεγονό ότι είμαστε ακόμα 500 εκατομμύρια πολίτες που συμμετέχουμε στην μεγαλύτερη ενιαία αγορά, στο μεγαλύτερο χώρο στον, ε, γεωγραφικό στον πλανήτη, στον οποίο μπορεί κανείς να ταξιδεύει ελεύθερα, ε, ξεχνούμε το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη τη παραμένουν οι πιο ανταγωνιστικέ οικονομίε στον κόσμο και ότι αυτέ οι χώρε είναι ελεύθερε και δημοκρατικέ. Τα ξεχνούμε όλα αυτά. Επομένω, θα πρέπει να ρωτήσουμε του εαυτού μα ποιε είναι οι επιλογέ που ανοίγονται μπροστά μα. Είναι προφανέ ότι όταν αλλάζει ο κόσμο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη θα πρέπει να αλλάξει. Όμω αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προβληματιστούμε προ ποια κατεύθυνση θέλουμε να αλλάξουμε, ποιο μέλλον επιθυμούμε για εμά και τα παιδιά μα. Προσωπικά ευελπιστώ ότι από αυτή την, περιοχή, αυτή την περίοδο της αβεβαιότητας θα περάσουμε σε μια περίοδο θάρρους. Ε, δηλαδή να, θα λαμβάνουμε με θάρρος τις αποφάσεις που χρειάζονται για να θωρακίσουμε την Ευρώπη και να την κάνουμε να αλλάξει προς το καλύτερο. Θα σας εκθέσω τις απόψει μου για το ποιε είναι οι πιο θεμελιώδει αλλαγέ, οι πιο ουσιαστικέ αλλαγέ, οι πιο ουσιαστικέ επιλογέ που ανοίγουν μπροστά μα και μετά θα έρθω στη λευκή βίβλο. Όσον αφορά τι θεμελιώδει επιλογέ, κατά την άποψή μου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει πιο ευέλικτη και να έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται με πολύ πιο γρήγορο τρόπο στι ε, αλλά υπάλληλε κρίσει. Και αυτή η ευελιξία σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνουμε αποφάσει πιο γρήγορα, να τι μεταβάλουμε πιο γρήγορα όταν χρειάζεται και να έχουμε τη δυνατότητα να κινητοποιούμε του πόρου που είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση των διαφόρων κρίσεων. Είμαι υπεύθυνη για την εκτέλεση του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχω ένα συγκεκριμένο μήνυμα να στείλω προ τα εθνικά κοινοβούλια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βοήθησε τα μάλα την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ε, έγινε η διαπραγμάτευση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρώπης. Και γιατί, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέμεινε να υπάρχει ευελιξία στην κατανομή των κονδυλίων του προπολογισμού. Και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα, την οποία την είχαμε πολύ μεγάλη ανάγκη, να τροποποιούμε την κατανομή των κονδυλίων εντός του προπολογισμού, όπως ανάλογα με το πώς χρειάζεται. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να βρούμε πόρους για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Αυτή τη στιγμή ε, έχουμε στη διάθεσή μα 16 δισεκατομμύρια, ενώ στην αρχή της κρίσης είχαμε 5. Αυτή η ευελιξία μας επέτρεψε να εστιάσουμε την δράση μας σε δύο προτεραιότητες που αφορούν τους πολίτες. Δύο, όχι είκοσι. Και οι δύο αυτές προτεραιότητες είναι η ανάπτυξη και η καταπολέμηση της ενεργείας αφενός και η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήματος ε, αφετέρου. Όταν μιλώ για ευελιξία, αντιλαμβάνομαι ότι η κατάσταση σημερινή απέχει πάρα πολύ από το ιδέατο. θα επιθυμούσα στο επόμενο ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη δυνατότητα μεταφοράς κοντιλίων για να αντιποκρινόμαστε στις αλλαγές. Ο κύριος Μάριο Μόντι, ο καλός μου φίλος, ο οποίος ασχολείται με τα ζητήματα των ιδίων πόρων, θα ε, ανέφερε επίσης το γεγονό ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο πώς ανακατανέμουμε τα έξοδα, αλλά πώς θα αυξηθούν και τα έσοδα. Για να θεωρηθεί επιτυχής η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταφέρνει να ανταποκρίνεται σε προβλήματα που είναι ουσιαστικά και μεγάλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αφουγκραζόμαστε τους πολίτες μας και να συζητάμε μαζί σας ποια θέματα θα πρέπει να λύνονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί αυτό είναι πιο αποτελεσματικό και ποια άλλα θέματα είναι καλύτερα να παραμένουν στο εθνικό. Αυτό σημαίνει λοιπόν μια δημοκρατική διαδικασία. Όχι όμως τόσο αργή και γραφειοκρατική όσο η δημοκρατική διαδικασία που έχουμε σήμερα. Τρίτο σημείο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε και εμείς. Και πιστεύω ότι αυτό θα το συζητήσετε και στη συζήτηση της έκθεσης της σχετικής. Τον Μάρτιο θα έχουμε τη Λευκή Βιβλίο στα χέρια μας, η οποία θα αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξελιχθεί στο μέλλον. Και όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επίσης και η ΟΝΕ. γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες ε, στην ε, συζήτηση αυτή. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, επιδιώξαμε να αποδείξουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα όταν χρειάζεται να λαμβάνουμε αποφάσεις γρήγορα και να τις υλοποιούμε γρήγορα και τα λέω γρήγορα, εννοώ με την ταχύτητα η οποία να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών. Παράδειγμα, η δημιουργία της συνοριοφυλακής και της ακτοφυλακής έγινε σε έξι μήνες. Ήδη λειτουργεί επιχειρησιακά. Σε όλα τα χρόνια που ασχολούμαι με τα ευρωπαϊκά, ποτέ δεν είδα μια απόφαση να λαμβάνεται τόσο γρήγορα και να υλοποιείται τόσο γρήγορα. Γιατί συμφώνησαν όλοι, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και κρατημέλη, ότι ήταν εξαιρετικά σημαντικό να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Γιατί ήταν απαραίτητο να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα για να μην ξεκινήσουν αυτές οι δημιουργίες εσωτερικών σύνορων που είχαν ξεκινήσει. Αντίστοιχη ταχύτητα θα έπρεπε να βρούμε και σε άλλα θέματα. Έτσι ώστε εν τέλει αυτό που είναι η εξαίρεση να γίνει ο κανόνας. Αυτή η ταχύτητα στη λήψη και την υλοποίηση της απόφασης. φαντάζομαι ότι θα συζητήσετε ε, τη της στην συνάντησή σα αυτή τον τρόπο με τον οποίο θα, θα εμπλέκονται περισσότερο στη λήψη αποφάσεων οι πολίτε. Γιατί όλοι διαπιστώσαμε δυστυχώ τα τελευταία χρόνια ότι όλο και περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται δακτυλοδεικτούμενη, ότι όλο και περισσότερα τα κράτη-μέλη, η πολιτική των κρατών μελών ε, κατηγορούν τις Βρυξέλλες και πολλέ φορέ συμβαίνει και το αντίθετο. Οι Βρυξέλλε να κατηγορούν ορισμένα κράτη-μέλη και αυτό το, αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει. Αυτέ οι αλληλοκατηγορίε δεν εξυπηρετούν. Γιατί ε, ε, έχουμε ένα ε, πλοίο το οποίο βρίσκεται στην, σε μια τρικυμία, βρισκόμαστε όλοι ε, στο ίδιο πλοίο, στην ίδια βάρκα, δεν έχει νόημα να ε, κατηγορούμε ο ένας τον άλλον για το τι έκανε και τι δεν έκανε. Βεβαίω είναι σημαντικά τα οικονομικά θέματα. Βεβαίω χρειαζόμαστε χρήματα για να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα. Όμω πολύ πιο σημαντικό είναι η ενότητα. Η ενότητα στο επίπεδο των θεσμικών οργάνων, η ενότητα στο επίπεδο των κρατών μελών, και η εν τέλει η ενότητα στο επίπεδο των ευρωπαϊκών λαών για να μην ε, βρισκόμαστε ε, ε, απέναντι σε αυτά τα προβλήματα που πολλοί πολίτες θεωρούν ότι δεν επιλύουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζετε ότι συνήθω δεν χειροκροτάμε. Ακούσατε όμω την αντίδραση και είμαστε πολύ ευγνώμονε. ο προπολογισμό είναι πάντα πολύ σημαντικό θέμα και δύσκολο. Νομίζω πάντως ότι θα είναι σημαντικό για όλους μας να δούμε πώς μπορούμε την Λευκή Βίβλο να τη μετατρέψουμε σε οδικό χάρτη και πώς ο οδικός χάρτης της Μπρατισλάβα ε, μαζί με τους άλλους οδικούς χάρτες ε, να μας ε, προχωρήσει στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας πω ότι αν θέλετε να παραμείνετε, μπορείτε να παραμείνετε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα προχωρήσουμε τότε στο πρώτο θέμα της Μεσσίας Διάταξης, που είναι το δικαίωμα εξετάσεις των πραγμάτων του Κοινοβουλίου. Και θα δώσω το λόγο στον ε, Ραμόν ε, Χαουρέκη. Αλλά όσο μιλάει, Μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο για να δούμε πόσο χρόνο μπορούμε να δώσουμε στον καθένα. Για μας ε, το θέμα αυτό ε, που είχε ξεκινήσει ήδη στο τέλος της προηγούμενης θητείας είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα από τα πιο δύσκολα θέματα διότι ακόμα και η διαδικασία που θεσπίζεται στη συνθήκη είναι πολύπλοκη. Και υπάρχουν αρκετά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα διάφορα θεσμικά όργανα, ιδιαίτερα το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Κάτι που αυξάνει τη δυσκολία που ούτως ή άλλως ε, υπάρχει με τον τρόπο διατύπωσης της συνθήκης. Το λέω αυτό Ε, για να μην επικεντρωθεί αποκλειστικά σε αυτό ώρα μόνο, ελπίζω να είναι επικοδομητικός στη σκέψη του. Αλλά τα τελευταία χρόνια είδαμε τις διαφορές αυτές ε, και γι' αυτό τώρα η Σλοβακική Προεδρία προσπαθεί να διευκολύνει την κατάσταση, κάτι που εκτιμούμε ιδιαίτερα. Απομένει όμως πολύς δρόμος ακόμα και θα ήθελα να καταλάβετε ότι υπάρχουν ε, διάφορες διαδικασίες, υπάρχουν κάποια προβλήματα στην ε, Ευρώπη που δεν ε, μπορούν να λυθούν αποκλειστικά με δράση στο υπερεθνικό επίπεδο, στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε λοιπόν κάποια θέματα κλειδιά, πάρα πολύ σημαντικά για τους πολίτες ε, και την άποψή τους. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτό το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων του Κοινοβουλίου για να συμβάλλουμε σε αυτό που κάνετε εσείς σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό για μας το θέμα αυτό και γι' αυτό αποτελεί και αντικείμενο της κοινή μας συζήτησης. Αυτά από μένα. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον Ραμόν Χαουρέγγι που είναι συγητής για αυτό το δύσκολο θέμα. Ραμόν, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα κυρία Επίτροπε, καλώς ορίσατε και να ευχαριστήσω και όλους εσάς εκπροσώπους των Εθνικών ε, Κοινοβουλίων. Η συζήτηση που μας φέρνει εδώ σήμερα για να συζητήσουμε μαζί σας απορρέει από ένα δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ε, επιτροπές ε, εξέτασης. Οι εξεταστικές επιτροπές, ε, όπως γνωρίζετε, είναι κατεξοχήν δικαίωμα των βουλευτών, διότι είναι στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα ευρύ φάσμα δικαιωμάτων προκειμένου να εξετάζει όταν υπάρχει κάποια δυναμία δικαίου ή όταν υπάρχει κάποια κακή εφαρμογή της νομοθεσίας ή κακή λειτουργία μέσω από πλευράς δημοσίων οργανισμών. Η συνθήκη της Λισαβόνας επέτρεψε ουσιαστικά ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και αυτά είναι και ένα από τα λίγα θέματα στα οποία το Κοινοβούλιο έχει νομοθετική πρωτοβουλία μαζί με τον εκλογικό νόμο που θα δούμε στη συνέχεια. Είναι ένα από τα λίγα πράγματα στα οποία έχει δικαίωμα πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, στα υπόλοιπα θέματα είμαστε εν αναμονή αυτών των οποίων προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όταν ξεκίνησε αυτή ε, η ε, εφαρμογή αυτού του δικαιώματος τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών αντιμετωπίσαμε ένα πολιτικό πρόβλημα πρώτη βαθμού διότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο στο οποίο ε, συμμετέχουν τα 28 κράτη-μέλη δεν συμφωνεί με τη σύσταση αυτών των επιτροπών και τα δικαιώματα τα οποία απορρέουν από αυτό και τις εξουσίες που μπορεί να έχουν αυτές οι εξεταστικές επιτροπές ε, για το Κοινοβούλιο. Σε μεγάλο βαθμό διότι υπάρχουν ε, σημεία ε, σύγκρουσης με τις εξουσίες των κρατών μελών, με τα εθνικά κοινοβούλια. Και παρά το γεγονός ότι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε έναν καρποφόρο θα έλεγα θετικό διάλογο, το Συμβούλιο περιορίζει ή αμφισβητεί τη δυνατότητα ε, πρωτοβουλίας ε, που θέλει ε, να πάρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να εξετάσει τα πράγματα. Να σας πω τώρα πού βρίσκονται τα προβλήματα, γιατί θέλουμε πραγματικά να ακούσουμε την άποψή σας. Έχουμε έρθει εδώ για να τίνουμε βίκο σε αυτά που έχετε να πείτε, διότι συνήθως το Συμβούλιο, όταν διαπραγματεύεται με το Κοινοβούλιο, μας λέει τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να έχετε εσείς αυτό το επίπεδο εξουσίας ε, εξέτασης. Πάντα βέβαια αναφερόμαστε στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά μπορεί να υπάρχει ε, κακή εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου ε, που να επηρεάζει ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη. Αυτό συνήθως συμβαίνει. Στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας μπορεί ε, τα κράτη να μην λειτουργούν αποτελεσματικά. Και επομένως η Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητά συγκεκριμένες δράσεις από ένα κράτος μέλος και εκεί μπορεί και να παρέμβει. Όταν λοιπόν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, για παράδειγμα, δικαίωμα η, Ευρωπαϊκή, ε, ε, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καλέσει ε, μέλη μια κυβέρνηση ενό κράτου μέλους ώστε να δώσουν πληροφορίε εδώ στην Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με κάποιο θέμα το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο ε, σύσταση μιας Εξεταστική Επιτροπής. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 12 του κανονισμού μας προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις στις οποίες ε, υπάρχει παραβίαση του δικαίου της Ένωσης ή κακοδιαχείριση όταν υπάρχουν και ευθύνε ενός οργάνου ή αρχής ενός κράτους μέλου, η Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορέσει να ζητήσει από το κοινοβούλιο του κράτους αυτού, από το Εθνικό Κοινοβούλιο, να συνεργαστεί στην εξέταση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε ίσως να συνάψει και διακοινοβουλευτικές συμφωνίες με τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Εδώ λοιπόν έρχεται και η πρώτη ερώτηση. Είναι λογικό κατά την άποψή σας ε, τα εθνικά κοινοβούλια να πρέπει να συνεργαστούν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν η εξέταση αφορά την ε, κακή διαχείριση ενός κράτους μέλους στην εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης. Αυτό, για παράδειγμα, είναι ένα από τα ερωτήματα τα οποία τίθενται. Στο άρθρο 13... La capacidad del Parlamento Europeo para indagar Ε, όταν υπάρχουν ερωτήσεις για την επικράτεια, ρωτάμε πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να είναι παρόν στη χώρα αυτή, όποια χώρα θέλετε εσείς, για να διερευνήσει επιτόπου κατά πόσον ε, επιτρέπεται, υπάρχει λόγος να γίνει επιθεώρηση. Και ε, αν θεωρείτε εσείς ότι υπάρχει δυνατότητα να επι παρέμβει. Στο 14 αναφέρονται οι, ε, τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα τεκμηρίωση. Το Ευρωπαϊ... Η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ζητήσει από τη χώρα, από το κράτος μέλος στο οποίο γίνεται η έρευνα, η εξέταση, ε, ή στα κράτη-μέλη, πιο συχνό είναι να είναι αρκετά τα κράτη-μέλη που εξετάζουμε, η εφαρμογή λοιπόν της νομοθεσίας στα κράτη-μέλη ε, ε, προβλέπει ότι θα πρέπει να δίνονται και αυτά τα έγγραφα. Και εδώ υπάρχει και μία σύγκρουση με το εθνικό δίκαιο, ώστε να μπορέσουν να επιτρέψουν την ε, προσκόμιση αυτών των πληροφοριών, ιδίω όταν αυτές οι πληροφορίες αφορούν εμπιστευτικά και τις πληροφορίες για το κράτος μέλος. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τους μάρτυρες. Η Εξεταστική Επιτροπή, σύμφωνα με αυτό το οποίο προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, μπορούμε να καλέσουμε οποιονδήποτε. Ευρωπαίο Μπορούμε λοιπόν να καλέσουμε οποιονδήποτε στην Εξεταστική Επιτροπή για να μας δώσει πληροφορίες. Είναι το άρθρο 15 το οποίο υποχρεώνει τον οποιονδήποτε από αυτούς να ε, ε, εμφανιστεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και πιο συγκεκριμένα η ε, Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διαβιβάσει το αίτημα στην Εθνική Αρμόδια Αρχή του κράτους μέλους όπου ε, βρίσκεται και εδρεύει το συγκεκριμένο άτομο και στα πλαίσια της ε, ε, δυνατότητες συνεργασίας και τις διατάξεις αυτές και ε, η αρχή της ε, χώρας μέλους θα καλέσει το εν λόγω άτομο να παρευρεθεί ενώπιον του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένως, η χώρα, η αρχή της χώρας είναι αυτή η οποία συγκαλεί το άτομο που θέλει να εξετάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα η Εξεταστική Επιτροπή να καλεί ε, υπαλλήλου ε, της κυβέρνησης ε, του κράτους μέλους, δημοσίου υπαλλήλου ή εκπροσώπους της κυβέρνησης, που η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να συγκολούνται για να δίνουν πληροφορίες. Βεβαίως, υπ' αυτή την έννοια, τίθεται και κάτι αντίστοιχο, διότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνεται η πρόσκληση από πλευρά κυβέρνηση του κράτους μέλους. Και τέλος όλα αυτά τελειώνουν με τη δυνατότητα πυθού που έχει η Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή ε, το να μπορεί να ασκήσει πιέσει ε, προς ε, ανθρώπους ή υπαλλήλους που καλούνται να παραστούν. Διότι εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων, λογικά αυτοί οι οποίοι καλούνται μπορούν κάλλιστα να μην μας δώσουν καμία σημασία. Όπως λοιπόν οι εξεταστικές επιτροπές των Εθνικών Κοινοβουλίων έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν κυρώσεις εάν κάποιος δεν είναι συνεργάσιμος και δεν ανταποκρίνεται σε μια πρόσκληση. Αντίστοιχα θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει ε, να απευθύνεται στην Εθνική Νομοθεσία και στο Κοινοβούλιο του κράτους μέλους για να ζητήσει ε, σε αυτή την περίπτωση να εφαρμόσει το αντίστοιχο καθεστώς επιβολής κυρώσεων και για αυτούς οι οποίοι δεν συνεργάζονται με τα αιτήματα της Ευρωεξεταστικής Επιτροπής. Αντίθετα, αντιλαμβάνεστε ότι κανεί δεν θα μας δώσει και φυσικά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και ένα πλαίσιο συνεργασίας με τα κράτη-μέλη, ώστε το σύστημα το οποίο έχει το κράτος μέλος προκειμένου να επιβάλλει αντίστοιχες κυρώσεις ε, όταν υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές, να είναι αυτό το οποίο θα δεχόταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς δεν ζητούμε ένα ξεχωριστό σύστημα ε, κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα και ξέρουμε ότι αυτό είναι δική σας αρμοδιότητα, αρμοδιότητα των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αλλά εάν ζητήσουμε στα πλαίσια της συνεργασίας ε, ε, μια εξεταστική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μπορεί να ζητήσει από ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη να επιβάλλουν αυτό το σύστημα, να εφαρμόσουν λοιπόν το σύστημα το οποίο προβλέπεται για τις εξεταστικές επιτροπές ε, στα δικά τους στα κοινοβούλια και να εφαρμόζεται και για την περίπτωση που η συνεργασία ζητείται από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τελείωσα κυρία Πρόεδρε. Κατ' ουσίαν αυτό το οποίο θέλουμε να έχουμε την άποψή σας. Διότι πολύ συχνά έχουμε την εντύπωση ότι το Συμβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί τους 28, όχι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά το Συμβούλιο έχει σοβαρές ενστάσεις ε, για την εφαρμογή ένας τέτοιου κανόνα από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, δεν μπορούμε να εγκρίνουμε τίποτα εάν δεν υπάρχει συμφωνία με το Συμβούλιο, διότι η συνθήκη της Λισαβόνας μας υποχρεώνει αυτός ο κανονισμός, αυτός ο ευρωπαϊκός νόμος που επιτρέπει τη ρύθμιση των εξεταστικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να την χάνει πρώτα τη σύμφωνη γνώμη ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Και το Συμβούλιο μας λέει τα κράτη-μέλη δεν είναι διατεθειμένα να δεχθούν αυτές τις εξουσίες ε, που μας δίνεται ως Κοινοβούλιο όσον αφορά τις εξεταστικές επιτροπές ε, που μπορεί να προκύψουν. Η κυρία Χούπνερ για παράδειγμα, είπε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο εξεταστικές επιτροπές, μία για τα Panama Papers και μία για το σκάνδαλο των εκπομπών της Volkswagen. Επομένως, ε, ε, εκεί κατά πάσα πιθανότητα υπήρχαν παράτυπες συμπεριφορές από πλευράς ευρωπαϊκών ή εθνικών αρχών στον έλεγχο των εκπομπών των οχημάτων. Επομένως, αυτή είναι η συζήτηση η οποία τίθεται και θα θέλαμε να ξέρουμε την άποψή σας. Αυτές είναι οι εξηγήσει ε, από πλευρά μου ε, κατόπιν υπόδειξης της Προέδρου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η, η, η Επίτροπος Γεωργίευα ε, αναγκαστήκε να φύγει, όμως έχουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις σχέσεις ε, με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, μεταξύ αυτών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βεβαίω και ο Γενικό Διευθυντή, λοιπόν, από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει το λόγο να μα εκθέσει τι απόψει του. Ε, έχω τέσσερα α, μέλη του, Ευρωπα... Ε, του Κοινοβουλίου στον κατάλογο ομιλητών. Δεν θα συνάγω από αυτό το ότι το ζήτημα δεν είναι ενδιαφέρον. Είναι γνωστό ότι πάντοτε στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χρειάζεται να τίθεται ένα χρονικό όριο στο χρονογόρευσης. Προσπαθήστε να το τηρήσετε αν είναι δυνατόν. Και θα ξεκινήσουμε από την κύριε Αζουμπάλη, Αντρώνης Αζουμπάλη από τη Λιθουανία. Έχετε το λόγο. Ε, ζητώ συγγνώμη κυρία Πρόεδρε γιατί ε, εγώ είχα ζητήσει το λόγο για το επόμενο θέμα συζήτησης. Ο κύριος Γιάννης Ντόσκι λοιπόν, μιας και έχουμε τρεις ομιλητές. Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα αυτό αναδεικνύει τα, τις θεσμικές ε, και συνταγματικές, συνταγματικά προβλήματα και συζητήσεις που διεξάγονται όχι μόνο στο ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά στο επίπεδο των κρατών μελών επίσης και πολλές φορές στο παρελθόν έχω, ε, ε, έχω εκφραστεί σε σχέση με τις αρμοδιότητες εξέτασης των πραγμάτων που αποδίδονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά την άποψή μου, επί της αρχής, θα έπρεπε κανείς να σέβεται την διάκριση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των υπολείπων εθνικών κοινοβουλίων. Από αυτή την έννοια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν διεξάγει εξεταστικές επιτροπές θα πρέπει να περιορίζεται στο, στις αποφάσεις και στις πράξεις των ευρωπαϊκών οργάνων και να αφήσει τον έλεγχο των εθνικών αρχών και των εθνικών κυβερνήσεων στα εθνικά κοινοβούλια. Ωστόσο αυτό είναι απλώς μια ιδανική περιγραφή των πραγμάτων. Ε, είναι δυνατόν να υπάρξουν αλληλοεπικαλύψεις. Ωστόσο, κατά την άποψή μου, αυτή η διάκριση αρμοδιοτήτων θα πρέπει να γίνεται σεβαστή. Βίως δεδομένου ότι η δημιουργία μιας εξεταστικής επιτροπής προσυδειάζει στην άσκηση ποινική δίωξη που θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε αυτό. Επομένω, δεν εκπλήσει το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα φιδωλό μέχρι στιγμή και δεν έχει εγκρίνει ε, τι προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι λογικό γιατί εκφράζεται εκεί η άποψη των κρατών μελών και ε, προστατεύονται τα συμφέροντα των κρατών μελών. Εάν το Ευρωπαϊκό Συνοβούλιο ε, περιοριστεί στις αρμοδιότητες του, πιστεύω ότι θα ήταν πιο εύκολο ε, να εγκρίνονται τέτοιες προτάσεις. Ο κύριος Άντιτς από την Ισπανία. Sí, <clears throat> muchas gracias. Bueno, en principio para eh, expresar que, que comparto el objetivo de, de... Καταρχάς να σας πω ότι συμφωνώ με το στόχο της έκθεσης ε, τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να συνεργάζονται με το δικαίωμα εξέταση των πραγμάτων της Ευρώπης και να υπάρχει καλύτερη ε, λογοδοσία για τα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Επομένως, ε, αυτό σίγουρα θα πρέπει να οδηγεί σε καλύτερη λειτουργία της διαχείρισης των ευρωπαϊκών πολιτικών και αυτά φυσικά σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε με ε, σαφήνεια τι ε, είναι αποτελεσματικό και τι αλλαγές χρειάζονται προκειμένου να αντιληφθούμε και να είμαστε σαφείς για το κατά πόσον ε, υπάρχει χρηστή διοίκηση. Εάν θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη φορολογική νομισματική ένωση και περισσότερες προσπάθειες για να καταφέρουμε τα πάντα από κοινού, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να διαθέτουμε κάποια κοινά απαραίτητα μέσα ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν όλα αυτά. Ε, ε, με την επιφύλαξη βεβαίως ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφής σεβασμός ε, για τις αρμοδιότητες οι οποίες είναι κοινέ και τις αρμοδιότητες του κάθε κοινοβουλίου. Σε κάποια θέματα υπάρχουν επικαλύψεις μεταξύ κάποιων πραγμάτων και επομένως αυτό το οποίο θεωρώ είναι ότι πρέπει να διαφυλάξουμε αυτές τις διαφορές και να υπάρχει συνεργασία με τα κράτη-μέλη και ε, να γίνονται τέτοιες συνεδριάσεις όπου ο καθένας θα μπορεί να ε, πει τις ιδέες του ε, για τα θέματα αυτά. Καταρχήν όμως να πω ότι υποστηρίζω τη συνεργασία προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ένας τρόπος να ενισχύσουμε τα κοινά, τα οποία κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ε, βλέπω κανέναν ε, βουλευτή να θέλει να πάρει το λόγο για το θέμα αυτό. Πρόκειται για μια διαδικασία όπου το Ευρωκοινοβούλιο χρειάζεται την ε, ε, συμφωνία και του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν είναι σημαντικός εταίρος στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά δεν θα ήθελα να χάσω την ευκαιρία αυτή η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωκοινοβούλιο. Ε, ίσως όμως λίγα λόγια να βοηθήσουν την όλη διαδικασία. Όσον αφορά το θέμα αυτό του δικαιώματος εξέταση ε, των πραγμάτων, νομίζω ότι έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για πρόοδο στο θέμα αυτό. Πρόκειται για έναν κανονισμό ο οποίος οδήγησε σε μια σειρά ε, ερευνών που ε, έδειξαν αφενός την επιτυχία του συστήματος, αφετέρου τις αδυναμίες, για παράδειγμα όσον αφορά την πρόσβαση σε έγγραφα. Υπάρχει επίσης ε, ανάγκη να εξυγχρονίσουμε τις διαδικασίες υπάρχει ανάγκη να εξυγχρονίσουμε τον κανονισμό αυτόν και όταν επικαιροποιεί κανείς έναν κανονισμό ε, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν. Πρώτον ένας διάλογος. Αυτό ε, είναι που συμβαίνει σήμερα και είναι πολύ χρήσιμος ο διάλογος αυτός. Επίσης, αν έχετε εκ των υστέρων τη δυνατότητα να μας υποβάλλετε τις παρατηρήσεις σας, ε, θα είναι πολύ χρήσιμο αυτό για να έχουμε μια εικόνα του πώς ε, οι εθνικές και ευρωπαϊκές ε, αρχές βλέπουν το θέμα. Υπάρχει όμως και ένα στοιχείο που προέκυψε κατά την προηγούμενη συζήτηση με τη Σλοβακική Προεδρία το να μάθουμε από τα λάθη μας. Έχουμε λοιπόν ε, πολύ, δύο πολύ σημαντικές επιτροπές εξέτασης ε, που δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή. Ε, η μία, η ΕΜΙΣ, θα εκδώσει σύντομα την σχετική της έκθεση, η άλλη επιτροπή αργότερα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε και αξιολόγηση των εργασιών. Όταν προτείνει κανείς έναν κανονισμό είναι πάντα χρήσιμο να γίνεται αξιολόγηση. Πάντως από τη δική μας πλευρά είναι σαφές ότι επικροτούμε την αναθεώρηση αυτή. Ήθελα να πω λίγα λόγια για τη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Μια συνεργασία που ξεκίνησε ιδιαίτερα μετά την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης. Ε, καταφέραμε να ε, επικοινωνήσουμε με σχεδόν ε, όλα τα κοινοβουλευτικά σώματα και πραγματοποιήσαμε σχεδόν 500 επισκέψεις στα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια από την αρχή αυτής της ηττίας. Δίνουμε μεγάλη σημασία στη συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια και νομίζω ότι και ε, το συγκεκριμένο θέμα θα είναι πολύ σημαντικό στη συνεργασία αυτή. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρωτού να δώσω το λόγο στον εισηγητή θα ήθελα να πω κάτι που ελπίζω να ε, εκλάβετε θετικά. Στο θέμα αυτό δεν προβλέπεται άμεσος ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων διότι είναι θέμα ε, διαθεσμικό σε με τον εκλογικό νόμο που υπάρχει εθνική διαδικασία για την ε, ε, έγκριση, την επικύρωση της νομοθεσίας. Εδώ πρόκειται για θέμα ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου με ειδική πλειοψηφία. Απαιτείται επίσης η συγκατάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ίσως όμως θα μπορούσαν τα εθνικά κοινοβούλια να στήσουν τη γνώμη των κυβερνήσεών τους σχετικά με τη θέση των κυβερνήσεων για το θέμα αυτό, διότι έχουμε κοινό συμφέρον με τα εθνικά κοινοβούλια να παράγουμε αποτελέσματα σε θέματα σημαντικά για τους πολίτες πολίτες που αναζητούν δίκαιη μεταχείριση και προσβλέπουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την αντιμετώπιση των θεμάτων που είναι σημαντικά για αυτούς. Σας έδωσα πριν το παράδειγμα των ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών ε, για την δίκαιη φορολόγηση, για τα έγγραφα του Παναμά κλπ. Πιστεύουμε λοιπόν ότι έχετε να παίξετε πολιτικό ρόλο. σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να στηρίξετε αυτές τις εξελίξεις όσον αφορά το ρόλο των κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δώσω το λόγο πάλι στον Ραμόν. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις απόψεις σας, παρόλο που δεν ήταν πολλές. Θα ήθελα να σταθώ σε τρία πράγματα τα οποία θεωρώ σημαντικά. Καταρχάς να επαναλάβω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας, και δεν είναι τυχαίο αυτό, έδωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να ρυθμίζει αυτό το δικαίωμα. Διότι εκφύσεως, ε, δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τη λαϊκή ε, κυριαρχία, διότι ξέρετε ότι μας εκλέγουν κάθε, ε, την ίδια μέρα σε όλη την Ευρώπη 500 εκατομμύρια πολίτες. Επομένως υπάρχει ένα στοιχείο πολιτικής νομιμοποίησης. Αυτή λοιπόν η δυνατότητα που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες σε ένα κοινοβούλιο συνδέεται με το δικαίωμα της εξέτασης όπως και όλα τα κοινοβούλια του κόσμου. Και δεν είναι τυχαίο το ότι η συνθήκη της Λισαβόνας ε, ακριβώς ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε το δικαίωμα να καθορίζει τον κανονισμό του. Πρώτο κρατούμενο αυτό. Δεύτερον, εμείς δεν πιστεύουμε και δεν δημιουργούμε ένα νέο ευρωπαϊκό δικαίωμα το οποίο να παραβιάζει οποιαδήποτε αρμοδιότητα οποιοδήποτε κράτους μέλους. Δεν δημιουργούμε ποινικό δίκαιο ε, δεν διανοούμαστε να πάμε τόσο πέρα πέρα, διότι το ποινικό δίκαιο είναι εθνική αρμοδιότητα. Δεν δημιουργούμε ένα σύστημα το οποίο να αποδυναμώνει τους κανόνες του κάθε Εθνικού Κοινοβουλίου σε θέματα εξέτασης. Σε καμία περίπτωση. Λέμε απλώς ότι όταν η δική μου έρευνα, η δική μου εξέταση φτάνει στη χώρα σου, το κοινοβουλευτικό σας σύστημα ή το ποινικό σας σύστημα ισχύει για αυτούς ή τους μάρτυρες ή τους υπαλλήλους που ε, θέλουμε να καλέσουμε. Και ε, προκειμένου να έχετε μια σαφή εικόνα του τι ακριβώς ε, διεκδικούμε. Πριν από λίγους μήνες στην Ευρώπη είχε ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Το σκάνδαλο των LuxLeaks. Μία χώρα ή περισσότερες χώρες, αρκετές χώρες, σίγουρα, μπορεί και πολλές, συμφωνώ, ασκούν μια φορολογική πολιτική την οποία θα μπορούσαμε ε, να θεωρήσουμε ότι είναι ε, ε, αθέμητη ενώπιον των γειτόνων τους. Προσφέρουν στις επιχειρήσεις τους ωφέλη για να εγκατασταθούν στη χώρα τους εις βάρος των συνεργατών τους ουσιαστικά, των άλλων χωρών. Και εγώ σας ρωτώ το εξής, δεν σας φαίνεται λογικό να το διερευνήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συστήσαμε μια επιτροπή. Αυτή τη φορά δεν ήταν εξεταστική επιτροπή, ήταν επιτροπή ενημέρωσης, την οποία αποκαλέσαμε Lux Leaks. Αντίστοιχο έχουμε κάνει τώρα με τα έγγραφα του Παναμά. Προς την ίδια κατεύθυνση πάμε. Έστω μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία την οποία εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη με τρόπο που δίνει δυνατότητα για απάτη. Έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαίωμα να διερευνήσει κατά πόσον η εφαρμογή μια γεωργική πολιτική, ενισχύσει κλπ. αποτελεί αντικείμενο απάτη σε κάποιε ε, κράτη-μέλη. Έχουμε δικαίωμα να τη διερευνήσουμε, ναι ή όχι. Έχουμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Το μόνο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι ποιες είναι οι εξουσίες ε, με τις, το οποίο συμφωνώ. Πρέπει να το συμφωνήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο ε, ώστε για παράδειγμα τα έγγραφα τα οποία ζητάμε αν είναι εμπιστευτικά, αν είναι απόρριτα του κράτους, ε, θα πρέπει να προστατεύονται δεόντως. Ή επίσης, εάν ένας μάρτυρας ζητήσει η κατάθεσή του να γίνει και κλεισμένο των θυρών, τότε να αναγνωρίζετε αυτό το δικαίωμα. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ρυθμίσουμε. Αλλά σας παρακαλώ δεν θα ήθελα να θεωρείτε ότι είναι συζητήσιμο το κατά πόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει ένα νόμο που να καθορίζει τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για εξέταση ε, των αδυναμιών εντό εισαγωγικών του ευρωπαϊκού δικαίου, όπου και αν εμφανίζονται. Διότι οι πολίτε θέλουν να ξέρουν εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανταποκρίνεται σε ένα σκάνδαλο σαν αυτό που σα ανέφερα προηγουμένω και θέλουν να γνωρίζουν κατά πόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσει μια απάντηση σε αυτό τον συναγερμό ώστε να μπορέσουμε να διορθώσουμε συμπεριφορές οι οποίες είτε μπορεί να είναι παράνομες είτε μπορεί να αποδυναμώνει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μας φέρνει εδώ και να σας ευχαριστήσω και πάλι για τη συνεργασία σας. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Διαπιστώνω ότι δεν έχει ζητήσει το λόγο κάποιος άλλος συνάδελφος για το θέμα. Μπορούμε να κλείσουμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη και να περάσουμε στο επόμενο, το δεύτερο της πρωινής μας συνεδρίασης, το οποίο είναι η συζήτηση για την αναθεώρηση του εκλογικού ε, δικαίου της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Θα κάνω εγώ την ε, εισήγηση την αρχική ως μία από τις εισηγήτριες, η δεύτερη είναι η κυρία Γιουλάινεν από τη Γερμανία και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν ήδη συνάδελφοι οι οποίοι έχουν ζητήσει το λόγο βεβαίως Όσοι ώρα κάνω την παρουσίασή μου έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε και το λόγο και να γραφείτε στον κατάλογο των ομιλητών χρησιμοποιώντα το ε, χαρτάκι που έχετε μπροστά σα. Όπως το δικαίωμα εξέταση, έτσι και το εκλογικό δίκαιο, ο εκλογικός νόμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία. Είναι, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, μια από τις λίγες διαδικασίες τις οποίες το δικαίωμα της πρωτοβουλίας επαφίεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως γνωρίζετε, κατά τα άλλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ουσιαστικά δεν έχει δικαίωμα πρωτοβουλίας. Είναι πολύ περιορισμένο αυτό στο τομέα της νομοθεσίας το άρθρο 223 στην πρώτη του παράγραφο της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι όσον αφορά το, Ευρωπαϊκό Εκλογικό Νόμο ε, η σύνταξη γίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γκρίνεται με ψηφοφορία στην Ολομέλεια με απλή πλειοψηφία. Κάτι το οποίο επίσης έχει συμβεί και μετά αποστέλλεται προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέρχεται ως πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τότε γίνεται η ψηφοφορία στην οποία απαιτείται η ειδική πλειοψηφία. Επομένως εκεί στο τέλος είναι της διαδικασίας που υπάρχει η μεγαλύτερη ασφαλιστική δικλίδα αν θέλετε. Και τέλος απαιτείται ανάλογα με τις συνταγματικές προϋποθέσεις και ρυθμίσεις σε κάθε χώρα μια διαδικασία επικύρωσης. Η διαδικασία λοιπόν αυτή όπως αντιλαμβάνεστε είναι ιδιαίτερως περίπλοκη και χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία από τη συνήθως μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί έχει δικαίωμα να υποβάλει παρατηρήσεις. Από την πλευρά μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βλέπουμε δύο πιθανές διαδικασίες, πι, ε, πιθανότητες. Θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε την ομοιόμορφη διαδικασία που προβλέπει η συνθήκη, δηλαδή μια διαδικασία η οποία θα είναι ίδια παντού, ανεξαρτήτως των εθνικών ιδιαιτεροτήτων και παραδόσεων, ή εναλλακτικά θα μπορούσαμε να θέσουμε κάποιες γενικές αρχές και έπειτα να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη, μεγαλύτερο περιθώριο ε, επιλογών. Επιλέξαμε την ε, πιο, τη δεύτερη διαδικασία, την πιο ευελίκτη διαδικασία. Και δυστυχώς όμως θεωρώ ότι αυτό δεν εκτιμήθηκε δεόντως στο επίπεδο των ε, κρατών μελών. Δηλαδή το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν προσπάθησε να επιβάλλει μια ομοιόμορφη διαδικασία. Ωστόσο, ταυτόχρονα προσπαθούμε να είμαστε ρεαλιστέ. Οι όποιε προτάσει μα να περιορίζονται μόνο στις απαραίτητα, στα απαραίτητα. Δηλαδή, μια επικυροποίηση της νομοθεσίας για τις ευρωεκλογές που η πιο πρόσφατη είναι από το 1976. Γνωρίζουμε πόσο έχει αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε και πόσο έχουν αλλάξει και οι προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίζει η Ένωση. Επίσης έχει αλλάξει και η σχέση των πολιτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο τρόπος με τον οποίο την ε, αντιμετωπίζουν. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντική και απαραίτητη η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου. Το έλεγε πριν και η Επίτροπο ε, Γεωργίευα, αλλάζει ο κόσμο, άρα πρέπει να αλλάξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο ισχύει και για την νομοθεσία η οποία ουσιαστικά ρυθμίζει την σχέση των πολιτών με, τη, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τα ευρωπαϊκά όργανα. Η νομοθεσία αυτή τη στιγμή ε, αφήνει μεγάλο περιθώριο επιλογών στα κράτη-μέλη για τον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσουν τι ευρωεκλογέ. Όμω θα θέλαμε να σταθούμε σε κάποιε βασικέ αρχέ, να διασφαλίσουμε κάποιε βασικέ αρχέ, έτσι ώστε στι ευρωεκλογέ του 2019 να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο για να έχουμε αυξημένη συμμετοχή των πολιτών και να αντιμετωπίσουμε πιο σοβαρά από ό,τι το έχουμε κάνει μέχρι στιγμή το λεγόμενο δημοκρατικό έλλειμμα. Έχουμε ε, καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες φαντάζομαι ε, θα έχετε εξετάσει. Και ο πρέσβης Γιαβόρτσικ της Σλοβακίας προηγουμένως έλεγε ότι και η Σλοβακική Προεδρία δίνει μεγάλη σημασία σε, στη συζήτηση που θα γίνεται. Ε, που γίνεται. Ε, στο επίπεδο των κρατών μελών για αυτήν την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είχαμε ξεκινήσει τη σχετική συζήτηση ήδη επί Λετωνική και Ολλανδικής Προεδρίας. Τώρα φτάσαμε πια στη Σλοβακική και η συζήτηση σίγουρα θα συνεχιστεί. Διαπιστώσαμε ότι η Σλοβακική Προεδρία από την πρώτη μέρα που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούλιο έδωσε σημασία στο θέμα. Έγιναν πολλές συναντήσεις με τις ομάδες εργασίας, και όπως ανέφερε και ο πρέσβης, αύριο θα συζητηθεί το θέμα στην Κορεπέρ στο επίπεδο των μονίμων αντιπροσώπων. Για πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο. Ε, όλα αυτά μας κάνουν να ευελπιστούμε ότι κατά τη διάρκεια της Μαλτέζικης Προεδρίας θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Θα γνωρίζετε εξάλλου ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη οι διαδικασίε για την επικύρωση του νομοθεσία για τι ευρωεκλογέ είναι και εκείνη χρονοβόρα, στο εθνικό επίπεδο χρονοβόρα. Επομένω πρέπει να βιαστούμε, πρέπει, πρέπει να κινηθούμε, εν πάση περιπτώσει, αρκετά γρήγορα, έτσι ώστε να μπορέσουμε οι ευρωεκλογέ του 2019 να διεξαχθούν με αυτή τη νέα νομοθεσία. Πριν να δώσω το λόγο στην συνάδελφο Γιολάινεν, θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Να αναφέρω ότι το θέμα αυτό έχει συζητηθεί και με τους ε, ε γενικούς γραμματείς των πολιτικών ομάδων στο Ευρωκοινοβούλιο και εκφράστηκε ε, στήριξη, πολιτική στήριξη στο να γίνει περισσότερο ορατά, περισσότερο ξεκάθαρα ε, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, να είναι ξεκάθαρο ότι είναι ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν στις ευρωεκλογές. Έτσι ώστε οι πολίτες που ψηφίζουν έναν ευρωβουλευτή να γνωρίζουν σε ποια πολιτική ομάδα θα ενταχθεί όταν πάει στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήταν λοιπόν ένα θέμα το οποίο ετέθη από αυτήν την πλευρά των θεσμικών οργάνων, αν θέλετε. Γιώ, είσαι έτοιμος να παρουσιάσεις την πρώτη. Uh, ναι, ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Νομίζω ότι το σημερινό είναι το κατάλληλο φόρουμ να μιλήσουμε για μεταρρύθμιση των ευρωεκλογών, του εκλογικού νόμου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν κοινή ευθύνη ώστε η έκκληση για συμμετοχή στους ε, ψηφοφόρους κατά τις ευρωεκλογές ε, να αποτελεί επιτυχία. Πρέπει να δείξουμε ότι οι εκλογές αυτές ε, είναι σημαντικές και να μην θεωρούνται εκλογές δευτέρας κατηγορίας. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι υπερβολικά σημαντικός για κάτι τέτοιο επειδή είναι νομοθέτης και νομοθετεί για κανόνες που ισχύουν για 500 εκατομμύρια ανθρώπους. Θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε προσπάθειες για να βελτιώσουμε τον τρόπο διεξαγωγής των ευρωεκλογών. Υπάρχουν κάποια ελλείμματα. Η κυρία Χίπνερ είπε ότι εργαζόμαστε με βάση εκλογικού νόμου από το 1976, πριν από 40 χρόνια. Ε, εγκρίθηκε αυτός ο εκλογικός νόμος, ο οποίος έχει εξελιχθεί ελάχιστα έκτοτε. Και βλέπουμε ότι κατά τις ευρωεκλογέ υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία πρέπει να ξεπεράσουμε. Και στους σκεπτικιστές ε, να πω ήδη από την αρχή ότι το θέμα δεν είναι ε, μόνο οι διαδικασίες. Ε, θα μου πούνε ότι το πρόβλημα είναι το περιεχόμενο, αλλά είναι σημαντικές και οι διαδικασίες. Έχουμε υποβάλει λοιπόν πρόταση που αποτελείται από διάφορα στοιχεία γνωρίζοντας ότι δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα θέματα εδώ ε, στον κύκλο μας διότι χρειαζόμαστε ομοφωνία ε, μεταξύ των 28 κρατών μελών στο Συμβούλιο. Και γνωρίζουμε ότι όταν απαιτείται ομοφωνία ε, ε, τελικά δεν περνούν οι μεγάλες ριζικές προτάσεις, ε, αλλά ε, βασιζόμαστε στον κοινό παρονομαστή. Ίσως σε μια επόμενη συνταγματική συνέλευση να πρέπει να κάνει τα μεγάλα βήματα. Είμαι ευγνώμων προ την Σλοβακική Προεδρία, διότι ήδη από την πρώτη μέρα, από την 1η Ιουλίου, την πρώτη μέρα που ανέλαβε την Προεδρία, έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό. και για το λόγο ότι ακόμα και ότι εάν δεν ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας μέχρι την πρωτοχρονιά, δεν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την πρόταση στις επόμενες ευρωεκλογέ ε, το 2019. Αλλά ήδη το 2018 θα αρχίσουμε να μιλάμε για τις ευρωεκλογέ ε, και θα λέει ο κόσμος ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ευχαριστώ λοιπόν ε, την Σλοβακική Προεδρία για τις προσπάθειές της ε, να βρει ε, τον κοινό παρονομαστή για την πρόταση. Έχουμε επιλέξει τρεις κατηγορίες ε, για τις βελτιώσεις. Η πρώτη κατηγορία είναι η διαφάνεια κατά την προετοιμασία των ευρωεκλογών. Υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, οι υποψήφοι επιλέγονται ήδη ένα χρόνο πριν. Ε, στη δική μου χώρα έξι με εννέα μήνες πριν γνωρίζουν οι υποψήφοι ότι είναι υποψήφοι και μπορούν να ξεκινήσουν την προεκλογική τους εκστρατεία. Ε, διότι οι εκλογικές περιφέρειες είναι στις περισσότερες χώρες μεγαλύτερες. Ενώ υπάρχουν άλλες χώρες όπου δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές δεν γνωρίζουν υποψήφοι ότι είναι υποψήφοι. Θέλουμε λοιπόν ε, ε, ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά ε, τους εκλογικούς καταλόγους, τα ψηφοδέλτια κλπ. Θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο λοιπόν όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα. Η κυρία Χίμπνερ επίσης είπε πολύ σωστά ότι μιλάμε για τις ευρωεκλογέ. Δεν έχουμε όμως ευρω... ευρωεκλογές, έχουμε 28 εθνικούς εκλογικούς νόμους 28 διαφορετικές προεκλογικές εκστρατείες, 28 διαφορετικά ψηφοδέλτια. Συχνά η Ευρώπη δεν συζητιέται καν κατά την προεκλογική εκστρατεία. Και στόχος ε, ήταν να κάνουμε τις ευρωεκλογές πιο ορατές, ε, τα κόμματα που ανήκουν σε κάποιο ευρωπαϊκό κόμμα να ε, χρησιμοποιούν το λογότυπο του, Ευρωπαϊκού Κόμματος ε, στα ψηφοδέλτια στη, κατά την ε, προεκλογική εκστρατεία. Διότι στο κάτω-κάτω οι περισσότεροι ε, ευρωβουλευτές ανήκουν σε κάποια ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια. Κάποιοι όχι, αλλά το 95% ναι. Και θα ήταν ένα πρώτο βήμα να δείξουμε αυτή τη σχέση που υπάρχει. Ευρωπαϊκά ψηφοδέλτια δεν ε, θα ε, έχουμε, είναι και αυτό μία πρότασή μας. Αντί για εθνικά ψηφοδέλτια να έχουμε ε, ευρωπαϊκά, αλλά αυτό μάλλον είναι ουτοπία. Η τρίτη κατηγορία, και θα ολοκληρώσω την παρουσίασή μου, είναι η ισότητα η ισότητα των ψήφων. Έχουμε δύο προτάσεις. Η μία αφορά την εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο Κοινοβούλιο. Στις συνθήκες έχουμε την αρχή μη διάκρισης ε, με βάση το φύλλο. Σε διάφορα κράτη-μέλη υπάρχουν διαδικασίες ε, για την εφαρμογή της αρχής αυτής ε, στις εκλογές. Και το δεύτερο θέμα είναι η ισότητα των ψήφων. 500 εκατομμύρια άνθρωποι είμαστε, 751 βουλευτές, όχι πολύ. Σε κάποιες χώρες με πολύ λίγες ψήφους αναλογικά ως προς ε, το, τον πληθυσμό ε, μπορεί να ε, λάβει κανείς έδρα του Κοινοβουλίου ενώ ε, σε άλλες χώρες ε, χρειάζονται πολύ περισσότερες ψήφοι και θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ισότητα, να υπάρχει δηλαδή ένα ελάχιστο κατόφλι και στα 28 κράτη-μέλη. Θα κλείσω εδώ. Τα υπόλοιπα στοιχεία της πρότασής μας ε, θα τα βρείτε στα έγγραφα. Θα χαρούμε αν ε, η Σλοβακική Προεδρία καταφέρει να θέσει το θέμα αυτό σε πολιτικό επίπεδο. Ίσως έτσι να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Και εσείς στα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια θα πρέπει επίσης να φροντίσετε για την εφαρμογή της πρότασης αυτής. Θα πρέπει να μας βοηθήσετε για να πετύχει αυτό. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Thank you. Ευχαριστώ αιτήματα. Άρα, μπορούμε να δώσουμε 5 λεπτά στον καθένα σας, ε, ακόμα και περισσότερο χρόνο αν χρειάζεστε. Δεν χρειάζεται να πιεστούμε και να σας περιορίσουμε. Ο κύριος ε, Σατζουβάλης καταρχάς λοιπόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί χρειαζόμαστε αναθεώρηση του εκλογικού νόμου. Υπάρχει πρόβλημα με την ε, δημοκρατική εκλογική διαδικασία στα κράτη-μέλη. Εγώ δεν έχω ακούσει για τέτοια προβλήματα, αλλά πολύ συχνά ακούμε ε, λογικά επιχειρήματα για την απόσταση μεταξύ της πραγματικότητας και τον τρόπο που την αντιλαμβάνονται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Επομένω, θεωρώ ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από μια κριτική αξιολόγηση αυτών των πραγμάτων. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω το ε, μότο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ενότητα στη διαφορετικότητα. Το να προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε ομοιομορφία σε όλα τα κράτη-μέλη είναι κατά της ποικιλομορφία ε, των παραδόσεων, των διαδικασιών και του ε, πολιτισμού των κρατών μελών. Επίσης πιστεύω ότι αυτή η ομοιομορφία θα οδηγήσει σε εκθετική ε, αύξηση των μικρότερων κομμάτων ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα θέσει κινδύνο πολιτικά κόμματα από τις μικρότερες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε πραγματικά λοιπόν να περάσουμε στην κυριαρχία δύο ή τριών πολιτικών οικογενειών και να μην υπάρχει εκπροσώπηση των ποικίλων ιδεών ε, που είναι ε, η ουσία της ευρωπαϊκής πολιτικής διαδικασίας. το να δείχνουμε το δημοκρατικό έλλειμμα και το κενό μεταξύ των ευρωπαϊκών ε, θεσμικών οργάνων είναι απαραίτητο, αλλά όχι με τρόπο που θα αποδυναμώνει περαιτέρω τα κράτη-μέλη και δεν θα σέβεται τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των τεχνητές αποφάσεις θα οδηγήσουν σε ένα νέο κύμα διαμαρτυριών και μόνο ε, πέραν των εθνικών ε, και κυρίως ε, πέραν του ευρωπαϊκού επίπεδου. Επομένως δεν υπάρχει λόγος για συζητήσεις εκλογικού νόμου χωρίς να υπάρχει υψηλότερο επίπεδο κυριαρχίας των κρατών μελών και χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις απόψεις των Ευρωπαίων πολιτών. Κύριε Πρόεδρε, τον Απρίλιο η Επιτροπή μας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μετά από διαβουλεύσεις ε, με άλλες αρμόδιες επιτροπές ε, και ε, πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο μας και με την κυβέρνηση γνωμοδότησε για τον προτινόμενο εκλογικό νόμο, την αναθεώρησή του και ξέρετε ότι ήταν μάλλον αρνητικές οι απόψεις στην καλύτερη περίπτωση ε, μετριοπαθής. Ο Ιστφαν Χόλινγκ από την Ουγγαρία τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να κάνω μια πολιτική παρατήρηση. Συμφωνώ με τον κύριο Γιώ Λάινεν που είπε ότι ελάχιστοι συμμετέχουν στις ευρωεκλογές. Πιστεύουμε ότι αυτό οφείλεται όχι τόσο στο γεγονός ότι δεν είναι σύγχρονος ο εκλογικός νόμος. Υπάρχουν βαθύτερα αίτια. Οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θέλουν να ψηφίσουν ε, γιατί δεν ε, τους ε, ικανοποιεί ο εκλογικός νόμος, αλλά γιατί δεν εμπιστεύονται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και πιστεύουμε ότι ο εξυγχρονισμός του εκλογικού νόμου δεν αρκεί για να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Πιστεύουμε ότι καλό θα ήταν να επανεξετάσουμε και πιθανόν να εξυγχρονίσουμε τον εκλογικό νόμο μεν, αλλά παρόλα αυτά θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα αρχής. Θεωρώ ότι η υποχρεωτική ψήφους ε, ε, θα σημαίνει ότι θα μπορούσε να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να αλλάξουν τον εκλογικό νόμο και να αλλάξουν τα όσα εφαρμόζουν. Δεν νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει. Δεν πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτές τις διατάξεις και τις συστάσεις. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να εφαρμοστεί αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά να σας πω ότι όσον αφορά τις εκλογές και την αναθεώρηση του εκλογικού νόμου θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Έχουμε αντίστοιχη ούτως ή άλλως νομοθεσία στην Ουγγαρία και μπορούμε να υποστηρίξουμε προτάσεις που αφορούν πολίτες που ζουν σε τρίτες χώρες για να μπορούν να ψηφίζουν και αυτοί ε, στις ευρωεκλογές. Όσον αφορά τις ε, προτάσεις όπως για παράδειγμα τη χρήση του λογότυπου των ε, πολιτικών ομάδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε υπέρ, αλλά να μην είναι υποχρεωτικό, να είναι απλώς σύσταση. Αν μπορέσουμε να κινηθούμε προς αυτή την κατάσταση, ε, θα μπορέσουμε ίσως να υποστηρίξουμε και την ε, πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ταϊάν Τζέιμς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λάινεν, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας σήμερα το πρωί. Μπορεί να εκπλήξει κάποιους ότι ως μέλος του Ηνωμένου Βασιλείου ε, μπορεί να θέλω και να σχολιάσω, διότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είμαστε στις ευρωεκλογές του 2019. Δεν υπάρχει όμως καμία εγγύηση. Επομένως θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις αν δεν σας πειράζει. Κύριε Λάινεν, στην έκθεσή σας, στη σελίδα 2, στην ενότητα 6, στο έγγραφο το οποίο μας δώσατε, ε, κάνετε πολύ ενδιαφέρουσε προτάσει. και θα ήθελα απλώ ε, να επισημάνω μια πτυχή που ενδιαφέρει όχι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη θεωρώ και πρέπει να τη λάβουμε υπόψη. Το πρώτο σχόλιο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι προτείνεται να υπάρχει μια κοινή προθεσμία 8 εβδομάδων πριν από τις εκλογές για ανταλλαγή δεδομένων και εγγραφή στα Μητρώα. Το Ηνωμένο Βασίλειο, παράδειγμα, ε, κάνει επαλήθευση των εκλογικών καταλόγων ε, το φθινόπωρο συνήθω ε, της προηγούμενη χρονιάς και αυτό επιτρέπει να ξεκινήσει μια πολύ καλή διαδικασία ώστε να μπορέσουμε να συλλέξουμε και να επαληθεύσουμε τα στοιχεία. Και δεν είναι κάτι το οποίο κάνουμε μόνο εμείς. Μήπως λοιπόν δεν αρκεί αυτό το διάστημα, κύριε Λάινεν, των 8 εβδομάδων και θα έπρεπε να το επανεξετάσουμε για να λάβουμε υπόψη όχι μόνο τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και άλλων χωρών και να διασφαλίσουμε ότι η ανταλλαγή των δεδομένων που γίνεται θα αντιμετωπίζει και την ε, πιθανότητα παράνομης εγγραφής και ε, παράνομης ε, ψήφου. Ε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι πρεσβείες στις άλλες χώρες χρησιμοποιούνται πάρα πολύ συχνά για εγγραφή και για ψηφοφορία. Και από ό,τι φαίνεται λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά. Επομένως, αν είναι ένα τμήμα μιας διαδικασίας που ούτως ή άλλως λειτουργεί αποτελεσματικά, γιατί να τα αλλάξουμε, γιατί να το πετάξουμε στα σκουπίδια. Η δεύτερη παρατήρηση είναι αυτό το δικαίωμα ψήφου στις ευρωεκλογέ για όλους τους πολίτες της Ένωσης που διαμένουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης φαντάζομαι το ερώτημα το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι ε, κατά πόσον έχει εξεταστεί επαρκούς το θέμα της ηθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε δει τι γίνεται με τους ε, ανθρώπους που έχουν διπλή ηθαγένεια και ζουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά έχουν και κάποια άλλη ηθαγένεια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε ένα κανόνα των 15 ετών που σημαίνει ότι όποιος ζει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να συμμετέχει. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή προσέγγιση. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε και αυτό, εάν δεν σας πειράζει, και να υπάρχει και μια, ένα κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Διότι υπάρχουν πολίτες που κάνουν συνειδητή επιλογή. Θέλουν να ζουν σε μια άλλη χώρα, εισφέρουν στην οικονομία εκεί, στον τρόπο ζωής εκεί. Γιατί λοιπόν να έχουν άποψη για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη-μέλη. Αντίστοιχα. Η τρίτη πτυχή δεν αφορά τόσο τον κατάλογό σας, αλλά την παράγραφο που έχουμε μετά από τον κατάλογο και αφορά το θέμα της εναρμόνισης της ελάχιστης ηλικίας ψήφου στα 16 χρόνια. Κατά την άποψή μου, και νομίζω ότι αυτό προέκυψε και στο δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ψηφοφορία είναι πάρα πολύ σημαντικό δικαίωμα και είναι και υποχρέωση, κάτι το οποίο υποστηρίζω απολύτω. Αλλά θα ήθελα να ε, παρατηρήσω το εξή. Αν οι νέοι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται τη φύση τη πολιτική, δεν αντιλαμβάνονται και τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν και αρχίζει να στρεβλώνεται αυτό το δικαίωμα και υποχρέωση ψήφου όσον αφορά την δική τους τη συνεισφορά. Θα ολοκληρώσω ε, αναφερόμενοι σε δύο σημεία που δεν είδα να καλύπτονται στην άκθεση. Γνωρίζω ότι υπάρχει πρόταση ε, υπό την προπόθεση ότι θα αποχωρήσει εγκαίρω το Ηνωμένο Βασίλειο πριν τις ευρωεκλογέ του 2019 για τη δημιουργία 73 εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για υπερεθνικά πολιτικά κόμματα. Μήπως θα μπορούσε ο κύριος Λάινε να το σχολιάσει αυτό το συγκεκριμένο για να δούμε κατά πόσον ε, θα μπορούσατε να το λάβετε υπόψη αυτό και αν έχετε γνωρίζετε αυτά τα σχόλια. Και υπάρχει και αυτή η πτυχή των εθνικών δημοψηφισμάτων. Η κυρία Χάρμς, η επικεφαλής των Πρασίνων, πριν από κάποιους μήνες ε, ζήτησε απαγόρευση αυτών των δημοψηφισμάτων. Τώρα ακούσαμε ακριβώ το ίδιο από τον κύριο Γιούντερ και τις προηγούμενες ημέρες. Έχω την αίσθηση ότι αν θέλουμε να συζητούμε εκλογές, αν θέλουμε να συζητούμε ψηφοφορίες, τότε σίγουρα πρέπει να ασχοληθούμε και με το θέμα των δημοψηφισμάτων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Άννα Μαρία Σούρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ πριν από 12 χρόνια ήρθα στην Ευρώπη ως μετανάστης και τώρα είμαι βουλευτής της Καταλωνίας ε, στο Κογκρέσο της Ισπανικής χώρας γιατί ε, το κόμμα μου θέλησε να προβάλλει το 20% του πληθυσμού ε, των μεταναστών που ζουν αυτή τη στιγμή στην Καταλωνία συμβιώνουμε εντός της περιοχής μας με έναν τρόπο που είναι συμβίωση για την ειρήνη και σεβόμενη τις διαφορές μας. Δεν πιστεύουμε ότι οι προκλήσεις ε, και η προσωμείωση των ανθρώπων σε άλλους πολιτισμούς είναι λύση. Πιστεύει ότι πρέπει να συμβιώνουμε και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό και σήμερα διεκδικώ και στην Ευρώπη το δικαίωμα ψήφου των μεταναστών. Καταρχάς, ε, διότι η ψήφος θα πρέπει να σχετίζεται και με την υπηκότητα ενός ανθρώπου και όχι ε, με την ηθαγένεια του, μόνο την εθνικότητά του. Και επομένως, ε, σε αυτή την Ευρώπη στην οποία συμμετέχουμε όλοι, πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή. Και επίσης γιατί θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος να περιορίσουμε αρκετά τα ρατσιστικά και ξενοφοβικά σχόλια τα οποία ανακύπτουν σε κάθε προεκλογική περίοδο και κατηγορούν ε, τους ανθρώπους για όλα τα κακά και τα δεινά της ανθρωπότητας γιατί δεν μπορούν να αντιποκριθούν στα μοντέλα τα οποία θεωρούν αυτοί ότι είναι σημαντικά και πρέπει να υπερασπιστούν. Δυστυχώ είδαμε αυτά τα οποία συνέβησαν στι Ηνωμένε Πολιτείε με τέτοιε ομιλίε σε προεκλογικέ εκστρατείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε ότι θα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και να περνά από τη θεωρία στην πράξη ε, για τέτοια θέματα που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα, ρατσισμό και ξενοφοβία. Πιστεύουμε ότι το δικαίωμα ψήφου θα βοηθήσει πάρα πολύ στην υλοποίηση αυτής της πρακτικής και κυρίως ε, θα επιτρέψει να συμμετέχουμε θετικά και δημοκρατικά όλοι οι πολίτες που και εμείς αποτελούμε τμήμα αυτής της νέας Ευρωπαϊκής Ένωσης του σήμερα, στην οποία θέλουμε να συμμετέχουμε προκειμένου να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλος για όλους. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε κυρία Σούρα. Ο κύριος Μαού από τη Γαλλία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να διευκρινίσω ότι αν και μεγαλόφωνος είμαι από το... Ε, προκατάγομαι από το Βέλγιο. Έχω κάποιες παρατηρήσεις για την πρόταση που μας υποβάλλεται υπάρχουν διατάξεις οι οποίες άπτονται της ορθής δημοκρατικής πρακτικής και αυτό πιστεύω ότι είναι σκόπιμο να το επενθυμίσουμε. Και γιατί να υπάρχουν εμπόδια για, την για τέτοιου τύπου προτάσεις ε, συνολικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, για την πρόταση να διασφαλίζεται η διαφάνεια στην, εκλογή, στην προεκλογική εκστρατεία, η ισοτιμία ή το ζήτημα του φύλου η ε, προστασία της ισότητας των φύλων. Όλα αυτά τα θέματα για εμένα είναι προφανή. Δεν βλέπω γιατί θα μπορούσαν να δημιουργούν προβλήματα οι επικλήσεις αυτών των αρχών. Θα ήθελα επίσης να επιθυμίσω ότι όλοι οι εκλεγμένοι ευρωβουλευτές εκπροσωπούν τον πληθυσμό που τους εξέλεξε, αλλά βεβαίως ε, αυτή η εκπροσώπηση γίνεται με κοινού κανόνες Ε, και αναφέρομαι για παράδειγμα στο ελάχιστο όριο, στο ελάχιστο ποσοστό. Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή διαβούλευση, συνένεση, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ποιο είναι το κατόφλι το οποίο θα πρέπει να ε, κανείς ξεπεράσει για να εκλεγεί. Τώρα, όσον αφορά τη συμμετοχή. Ευτυχώς η χώρα μου συνεχίζει να είναι εξαίρεση. Σε εμά είναι υποχρεωτική η ψήφος. Επομένως, ε, το ζήτημα της συμμετοχής τίθεται πολύ λιγότερο από ό,τι σε κάποια άλλα κράτη-μέλη. Ίσως είναι και αυτός ένας τρόπος για να ευαισθητοποιήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες για τα θέματα, τα, τα κοινά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένοι ανέφεραν την ψήφο Ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται στο εξωτερικό. Ε, πιστεύω ότι είναι το ζήτημα σημαντικό, γιατί δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί και εντό παρεθέσεως να υπενθυμίσω ότι οι ευρωεκλογέ ε, σε κάποιες χώρες ε, ε, συνδέονται με άλλες εκλογές. Δύσκολα μπορεί να φανταστεί λοιπόν κανείς μια εκλογική διαδικασία στην οποία θα υπάρχουν διαφορετικά εκλογικά σώματα ανάλογα με το σε ποια εκλογή κανείς συμμετέχει. Επομένως θα πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας σε μια προσπάθεια εναρμόνισης. Τώρα, όσον αφορά τη μείωση του ορίου ηλικίας ε, στα 16 έτη. Δεδομένου ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν ε, εγκρίνει κάτι τέτοιο, δεν έχουν υιοθετήσει κάτι τέτοιο για τις δικές τους εθνικές εκλογές, θα μου φαινόταν παράλογο ε, να υπάρχει ένα διαφορετικό ελάχιστο όριο ηλικίας για τις ευρωεκλογέ από ότι για τις εθνικές εκλογές. Δύσκολα κανείς θα μπορούσε να εξηγήσει αυτό, αυτή την επιλογή. Να σας πω εν είδη ανεκδότου ιστορίας ότι γνωρίζω οι συμπολίτε μα οι οποίοι έχοντα διπλή υπηκότητα, κατάφεραν να ψηφίσουν δύο φορέ στις δύο χώρε του επειδή τυχαίνει να είναι και γειτονικέ και να εύκολο να περάσει κανεί από τη μια στην άλλη, ε, δύο φορέ στις ευρωεκλογέ. Επομένω, το ζήτημα του ελέγχου των εκλογικών καταλάνων λόγων είναι υπαρκτό και θα πρέπει να φροντίσουμε να το ρυθμίσουμε γιατί μπορεί να, ε, υπάρξουν, ε, να επηρεάσει αυτό το, το, τέτοιου τύπου απάτες στο τελικό αποτέλεσμα. Επομένως, θα έλεγα ότι τα θέματα αυτά ήδη συζητώνται, συζητώνται στο Βέλγιο, σε άλλες χώρες. Ε, το ζήτημα της ε, ε, ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θέτει το ζήτημα αυτό. Ακόμα περισσότερο εάν συζητήσουμε την πιθανότητα να υποβάλλονται ψηφοδέλτια μέσω του ίντερνετ, εκεί πραγματικά θέτει το, το ζήτημα της ασφάλειας της ψηφοφορίας. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει πολύ ευρύτατη διαβούλευση διαδεδομένων των διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στα, στα διάφορα κράτη-μέλη. Ωστόσο, όπως είπα και στην αρχή, δεν βλέπω γιατί να υπάρχει οποιαδήποτε αντίρρηση στο να υπάρχει μια επενθύμηση γενικών αρχών και βέλτιστων πρακτικών. Εντό ενό γενικού πλαισίου, λοιπόν, να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα κρατών μελών συγκεκριμένα. Ευχαριστώ, Γιάννα Κλασοπρανσκή. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι το ερώτημα κλειδί στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουμε είναι η αιτία για την ε, χαμηλή συμμετοχή στις ευρωεκλογέ. Νομίζω ότι οι πολίτες μας ε, θεωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση οντότητα απομακρυσμένη από τα τοπικά προβλήματα των κρατών μελών. Άσχετα από το ποια είναι η πραγματικότητα, έτσι αντιλαμβάνονται οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τρόπος που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σύστημα της κίτρινης κάρτας. Είναι κάτι που είναι δύσκολο να γίνει στα εθνικά κοινοβούλια όταν απορρίπτουμε λοιπόν την κίτρινη κάρτα θα πρέπει να επιδεικνύουμε περισσότερο σεβασμό στις εργασίες των εθνικών κοινοβουλίων. Επίσης, ε, ε, άμεσες ε, εκλογές για την εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, αυτή λοιπόν η αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο απομακρυσμένη οδηγεί σε χαμηλή συμμετοχή σε ευρωεκλογέ και χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η συμμετοχή στις εκλογές ε, έχει έμεσες συνέπειες ε, στην πολιτική. Η άμεση εκλογή του Προέδρου του Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, θα αυξήσει πιθανότατα την συμμετοχή στι εκλογές, θα συμβάλλει όμω σε περισσότερες εξουσίες ε, για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ίσως αυτόν τον δρόμο θα έπρεπε να επιλέξουμε στο μέλλον. Υπό το φως όμως του ευρωσκεπτικισμού που επικρατεί, μια τέτοια λύση θα ήταν αντιπαραγωγική και θα οδηγούσε στην υπονόμευση της Ευρωπαϊκής Συνοχής. Όσον αφορά την εναρμόνιση του χρονοδιαγράμματος των ευρωεκλογών με τις ε, προθεσμίες για την εκπόνηση των εκλογικών ε, καταλόγων, ε, την ψήφο από το εξωτερικό ή τα λογότυπα των ευρωπαϊκών κομμάτων είναι προτάσεις τις οποίες μπορούμε να εξετάσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σύνθημα το ενωμένη στην πολυμορφία και θα ήταν χρήσιμο ε, να μην είμαστε αντιεπικοδομητικοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Χρύμπνερ που μας προσκαλέσατε σήμερα εδώ και που θέσατε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη και που μας θυμήσατε πόσο ιδιαίτερη είναι η νομοθετική διαδικασία στο θέμα αυτό. Το Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου εκτιμά ότι το Κοινοβούλιο δεν επέλεξε ενιαία διαδικασία παντού, αψηφώντας ε, τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Ε, από την άλλη, συμφωνούμε ότι μετά από 40 χρόνια πρέπει να συζητήσουμε τροποποίησεις ε, του, της νομοθεσίας, δεν θα έλεγα αλλαγές, αλλά προσαρμογές της νομοθεσίας. Για μένα προσωπικά είναι ενδιαφέρουσα και σημαντική η ορατότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Ε, γνωρίζω όμως ότι σε κάποιες χώρες, σε κάποια κόμματα, ε, πάνω από ένα κόμματα ανήκουν στην ίδια πολιτική ομάδα εδώ, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα. Επίσης, ε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ο ε, κύριος Λάινεν ανέφερε ότι η ισότητα των φύλων είναι ε, σημαντικό θέμα και την προηγούμενη εβδομάδα στο κοινοβούλιο μας ε, ψηφίσαμε πρόταση που έλεγε ότι οι υποψήφοι θα πρέπει να είναι κατά 50% άντρες και κατά 50% γυναίκες στις εκλογές. Έτσι θα πετύχουμε καλύτερη εκπροσώπηση των δύο φύλων. Επιτρέψτε μου να θέσω μια ερώτηση θα με ενδιέφερε η συζήτηση σχετικά με τον κορυφαίο υποψήφιο. Φαντάζομαι ότι το Συμβούλιο δεν το βλέπει πολύ θετικά αυτό. Οι συζητήσεις εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λοιπόν, τι δείχνουν όσον αφορά αυτή την έννοια. Ευχαριστώ. Α, και να προσθέσω Στη χώρα μου είναι σημαντικό και το θέμα των πολλαπλών ψήφων. Έχουμε πολλούς πολίτες που είναι υπήκοοι ε, πάνω από ενό κράτου μέλου. Ε, αρκετοί φίλοι που είπαν ότι έχουν ψηφίσει ε, πάνω από μία φορά. Νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα και να το ελέγξουμε καλύτερα. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τελμίρα Μπαρέιρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Όσον αφορά το θέμα αυτό, συζητήθηκε και πολλές από τις παρεμβάσεις που ακούσαμε εδώ ε, με αυτό ασχολήθηκαν. Είδαμε ποια είναι τα αίτια αυτής της χαμηλής συμμετοχής στις ευρωεκλογέ. Ε, εάν δεν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε προς τα αίτια, πολύ πιο δύσκολα θα συμφωνήσουμε προς τις λύσεις. Ε, ένα κόμμα σαν το δικό μου ή πολλά ε, από εκείνους που μίλησαν πριν, ε, ως ευρωπαϊστές πρέπει να συμφωνήσουμε για την ανάγκη να ενισχύσουμε την νομιμοποίηση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και να βελτιώσουμε την δημοκρατική σχέση και την προβολή των κομμάτων ε, και των ευρωεκλογών. Και φυσικά υπάρχουν διαφορετικοί όροι και σίγουρα από πλευρά τη χώρα μου πρέπει να τα θέσουμε και στο σωστό πλαίσιο. Διότι πολλά από αυτά τα οποία προτάθηκαν εδώ σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταρρύθμισουμε γενικότερα το εκλογικό καθεστώ και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να είναι πρωτοβουλία ενό κόμματο και δεν μπορεί να είναι και μονομένη πρωτοβουλία τη κυβέρνηση. Ε, σε γενικές γραμμές ε, γίνεται τροποποίηση με ευρεία συνένεση όπως θα πρέπει να είναι διότι αυτό είναι ένας από τους βασικούς κανόνες του δημοκρατικού μας συστήματος. Πρόσφατα εγκρίθηκε μια τροποποίηση του εκλογικού νόμου για μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ε, και υπήρχε πολύ μεγάλη συνένεση από αυτού και πριν από λίγες εβδομάδες ε, λήφθη υπόψη και άλλη τροποποίηση προκειμένου να μειωθεί η ηλικία συμμετοχή στις εκλογές ε, στην οποία όμως δεν υπήρχε συμφωνία, υπήρχε μια κάποια διαίρεση στο Κοινοβούλιο και σε μια χώρα όπου ο εκλογικός νόμος και οι εκλογικοί κανόνες απαιτούν μεγάλη συνένεση και πρωτοβουλία Κοινοβουλίου από πολλές πλευρές σημαίνει ότι τουλάχιστον στην Ισπανία οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να τύχει ε, ενδελεχούς εξέτασης και θα πρέπει να την χάνει και ευρύτατη της υποστήριξης. Ευχαριστώ πολύ. Ah, uh, Madame η κυρία Ιπνερ έφυγε, προεδρεύω εγώ για λίγο. Η κυρία Τριανταφύλου. Δεν ξέρω αν πρόφερα σωστά το όνομά σας. Πρέπει να φύγετε, οπότε σας δίνουμε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σωστά το προφέρατε. Καλημέρα σε όλους. Είναι πραγματικά ένα σημαντικό ζήτημα, όχι αυτό καθ' αυτό ένας εκλογικός νόμος, αλλά είναι σημαντική η συζήτηση για τον τρόπο αλλά και το εύρος της συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, γιατί συζητάμε σήμερα για την αλλαγή της εκλογικής διαδικασίας του εκλογικού νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί σήμερα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει την εντύπωση ότι βρίσκεται υπό εκαθάριση ή στην καλύτερη περίπτωση βιώνει εξαιρετικά μεγάλους κλειδονισμούς. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι εκλογικοί νόμοι προάγουν εκλογικά αποτελέσματα όχι τόσο με την έννοια των ποσοστών, των ποσοτικών αποτελεσμάτων, αλλά προάγουν πολιτικό αποτέλεσμα. Και επομένως θα πρέπει πάντοτε η πολιτεία και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να προκρίνει εκείνες τις διαδικασίες και να θεσπίζει εκείνους τους νόμους όχι μόνο για την καλύτερη συμμετοχή αλλά και την ίση δυνατότητα για συμμετοχή. Στις προτάσεις που διάβασα υπήρχαν ε, αρκετές προτάσεις που έχουν ενδιαφέρον. Νομίζω ότι η προσπάθειά μας για τεχνικές έτσι βελτιώσεις δεν θα έχουν πάντοτε διαφοροποιήσεις. Μπορούμε δηλαδή σε κάποια σημεία να συμφωνήσουμε. Νομίζω όμως ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε ότι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν άλλα προβλήματα. Μίλησαν όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές για τη μικρή συμμετοχή στις ευρωεκλογές. Δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις, ούτε τυπικές. Δηλαδή, ωραία, το προσπερνάμε και πάμε να δούμε με ποιες αλλαγές τεχνικές θα βελτιώσουμε τη συμμετοχή, θα αυξήσουμε τη συμμετοχή. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει με μεγάλη γενναιότητα να αξιολογήσουμε και τον εκλογικό νόμο και τον την εκλογική διαδικασία στις ευρωεκλογές, αλλά πάνω από όλα νομίζω ότι ήρθε η στιγμή ως Ευρωπαίοι πολίτες που θέλουμε να συνεχίσουμε μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια να αξιολογήσουμε τα πεπραγμένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν είναι εύκολο. Και δεν μιλώ μόνο για τις πολλές και μεγάλες διαδικασίες ε, τις νομοθετικές που χρειάζονται και τις αλλαγές, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και για το προσφυγικό και για το μεταναστευτικό. Θα έχουμε φεύγει τη δυνατότητα όταν μιλάμε για το μέλλον της Ευρώπης, το άλλο θέμα, να πούμε δύο πράγματα και γι' αυτό. Δεν αρνιέται κανείς την καθολικότητα της ψήφου, δεν αρνιέται κανείς τη διαφάνεια, δεν αρνιέται κανείς την ισοτιμία, δεν αρνιέται κανείς τις βιλτιώσεις σε σχέση με την ισότητα των δύο φύλων, αλλά μιας και μιλάμε ας πούμε γι' αυτό, ας το πάρω ως παράδειγμα. Ας δούμε τι συμβαίνει στις γυναίκες ακόμα και στο δυτικό κόσμο. Νομίζω ότι περισσότεροι από εδώ μέσα γνωρίζετε ότι η πρώτη αιτία θανάτου γυναικών, ακόμα και στη Δύση, δεν είναι ο καρκίνος ή κάποια αρρώστια, αλλά είναι η βία από τους συντρόφους τους. Επομένως το λέω αυτό για να πω ότι μια τεχνική έτσι ε, πρόταση δεν μπορεί να λύσει άλλα ζητήματα που είναι αμυγός πολιτικά. Θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη συμμετοχής και ειλικρινούς διαλόγου και θεωρώ ότι θα πρέπει να πάμε στο δρόμο της συνευθύνης, να βαδίσουμε το δρόμο ως Ευρωπαίοι πολίτες της συνευθύνης και όχι της ετεροπιθαρχίας. Από αυτή τη γενική αρχή νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε και ως προς τις τεχνικές λεπτομέρειες, αν πραγματικά μας ενδιαφέρει η ισοτιμία, αν πραγματικά μας ενδιαφέρει οι ευρωπαϊκές χώρες να λειτουργούν ισότιμα και τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα κράτη, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν άλλες αλλαγές, πραγματικές, ουσιαστικές και πολιτικές αλλαγές και να συζητήσουμε εκ των υστέρων τις αλλαγές, τις τεχνικές, γιατί δεν είναι τεχνικές αυτές οι αλλαγές που προτείνονται εδώ, δεν είναι ουσιαστικές πολιτικές. Σας ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εκπροσωπώ την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Πολωνίας. Έχουμε υποβάλει έγγραφα με πολύ αρνητικές θέσεις ε, σχετικά με την πρόταση. 20 βουλευτές υπερψήφισαν αυτή την επικριτική γνωμοδότηση. Μόνο μία αντίθετη ψήφος υπήρχε. Πράγμα που δείχνει ότι στο Πολωνικό Κοινοβούλιο και το κυβερνών κόμμα και μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης συμμερίζονται τη θέση αυτή. Ε, το πρόβλημα δεν είναι ο εκλογικός νόμος σύμφωνα με τον οποίο διεξάγονται οι ευρωεκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο δημοψήφισμα για το Brexit. Η συμμετοχή στις, ε, στο δημοψήφισμα ήταν ε, πολύ ψηλή, σχεδόν 70%. Ε, οι κανόνες οδήγησαν σε τόσο μεγάλη συμμετοχή. Όχι, το θέμα ήταν τόσο σημαντικό. Φοβάμαι ότι οι ευρωεκλογέ ε, δεν προσελκύουν το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με θέματα που ελάχιστα ενδιαφέρουν τους πολίτες. Ωστόσο, Μάλλον οι ε, ε, ε, ευρωπαίοι πολιτικοί ασχολούνται με θέματα τα οποία ελάχιστα ενδιαφέρουν τους ευρωπαίους πολίτες. Το θέμα λοιπόν δεν είναι το λογότυπο των ευρωπαϊκών κομμάτων ή τα κοινά εκλογικά πρότυπα, ούτε η προθεσμία για την πρόταση των υποψηφίων στα κράτη-μέλη. Τα θέματα αυτά δεν θα επηρεάσουν την συμμετοχή των ψηφοφόρων. Ας ασχοληθούμε λοιπόν με τα βασικά προβλήματα της Ευρώπης για να έχουμε υψηλή συμμετοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει κανείς άλλος που να θέλει να πάρει το λόγο, διότι κλείνουμε αυτό το μέρος της συζήτηση. Υπάρχει κάποιο ευρωβουλευτής που θα ήθελε να αναφερθεί ε, στον εκλογικό νόμο. Όχι, δεν θέλει κανεί το λόγο, οπότε μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτηση. Θα ολοκληρώσουμε λοιπόν τη συζήτηση. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον Γιώ και μετά θα πάρω και εγώ το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για τις απόψεις σας, τις παρατηρήσεις σας. Είναι σημαντικό για μας να ακούσουμε τις ε, απόψεις στα Εθνικά Κοινοβούλια. Ε, είπα ήδη από την αρχή ότι ο καλός εκλογικός νόμος δεν μπορεί να υποκαταστήσει την καλή πολιτική. Ε, πολλοί είπαν γιατί ασχολούμαστε με τον εκλογικό νόμο τη στιγμή που έχουμε ένα σωρό άλλα προβλήματα όπως είναι η μετανάστευση, η οικονομική κρίση ε, κλπ. Δεν νομίζω ότι είναι ε, δίκαιο να χρησιμοποιούμε το ένα εις βάρος του άλλου. Χρειαζόμαστε και τα δύο. Χρειαζόμαστε καλή πολιτική, χρειαζόμαστε όμως και καλή δημοκρατική πρακτική, όπως είπε ο συνάδελφος Μαό από το Βέλιο. Θέλουμε λοιπόν καλή δημοκρατική πρακτική ε, για τις κοινέ μας εκλογές ενός ε, κοινοβουλευτικού, κοινού, ε, κοινού κοινοβουλευτικού σώματος. για τους βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια όπως και για τους πολίτες σημαντικά είναι τα προβλήματα και όχι με σύμφωνα με ποιου κανόνε θα συμμετάσχω στι ευρωεκλογέ ε, το 2019, αλλά να το χρησιμοποιούμε αυτό ως επιχείρημα δεν είναι σοβαρό. Θέλουμε και στις χώρες μας να έχουμε καλό εκλογικό νόμο, διότι καλούμε τους πολίτες μας να συμμετάσχουν σε αυτήν ε, την ε, δημοκρατική δραστηριότητα. Και με την νομοθεσία, με τους κανόνες που θεσπίζουμε, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, που συνερχόμαστε στο Στρασβούργο από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Θεσπίζουμε κανόνες πολλούς για την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλούμε τους πολίτες να εκλέξουν τους ανθρώπους που μπορούν να τους εκπροσωπήσουν καλύτερα κατά τη θέσπιση αυτών των κανόνων. Και επειδή είμαστε μια ανοιχτή φιλελεύθερη ε, δημοκρατία, ακόμα λέω εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι βλέπω διάφορες ε, τάση κέντρο Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μη δημοκρατικές, σε κάτι που μου προκαλεί πονοκεφάλους ε, το να σκέφτομαι τι μπορεί να μας συμβεί στο μέλλον. Οι πολίτες ε, λοιπόν έχουν τη δυνατότητα και κατά τις προεκλογές ε, να ρίξουν ψήφο διαμαρτυρίας. Όλα αυτά είναι θεμητά. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι κάποιες από τις παρατηρήσεις σας έδειξαν ότι μπορούμε να προσαρμόσουμε το σύστημα, όπως είπε ο κ. Σέγγελ. Διότι εφαρμόζουμε ακόμα τον εκλογικό νόμο του 1976. Όποιος θέλει να παραμείνει στον προηγούμενο αιώνα, ας το κάνει. Εγώ όμως δεν θέλω να κολλήσω στον προηγούμενο αιώνα. Θέλω ε, να συνοδεύσω και να ακολουθήσω τις εξελίξεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι ε, έτσι απάντησα σε μια σειρά παρατηρήσεων που έλεγαν ότι δεν είναι σημαντικός ο εκλογικός νόμος. Για μένα είναι κάπως επιφανειακό αυτό το επιχείρημα. να πω στον κύριο Τσουμπάλης και σε άλλους, δεν εναρμονίζουμε τον Ευρωπαϊκό Εκλογικό Νόμο, προσπαθούμε να βρούμε κοινούς κανόνες για την καλή δημοκρατική πρακτική. Ε, ήταν πολύ ωραία η διατύπωσή σας. Και σε πολλούς τομείς Έχουμε ελάχιστα πρότυπα όπως για την προστασία του περιβάλλοντος, για την προστασία του καταναλωτή. Επιδιώκουμε να έχουμε ελάχιστα πρότυπα και σε άλλους τομείς. Έχουμε κοινά πρότυπα και για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Έχουμε επίσης το καθεστώς των ευρωβουλευτών. Ε, δεν έχουμε όμως ε, καθεστώς, δεν έχουμε κοινά πρότυπα για τις ευρωεκλογέ, ε, το οποίο είναι πολύ περίεργο. Απομένει πολύ ο δρόμος για μας, διότι έχουμε μείνει με την εκλογική πράξη του 1976. Δεν εναρμονίζουμε Θέλουμε όμως να κάνουμε κάποιες προσαρμογές ε, για να προσαρμοστούμε σε κάποιες γενικές αρχές που έχουμε διατυπώσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτό απαντάει και στην παρατήρηση του κυρίου Ανσουμπάλης και αναφέρατε το σύνθημα ενωμένη στην πολυμορφία. δεν μπορούμε να εναρμονίσουμε τις ε, προεκλογικές εκστρατείε, ε, διότι είναι διαφορετική η κουλτούρα σε κάθε κράτος μέλος. Ε, θέλουμε όμως να έχουμε κάποια ελάχιστα πρότυπα. Κύριε Γόλιτς, είπατε ότι δεν θέλετε υποχρεωτικούς κανόνες όλοι να είναι προαιρετικοί. Καλώς, μείνει και αυτό μια άποψη. Εντός η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και μια κοινότητα κανόνων και δικαίου. Και μερικές φορές είναι χρήσιμο να έχουμε κοινούς κανόνες ε, για να επικρατούν κοινέ ε, συνθήκες. Και κατά τις ευρωεκλογές οι ευρωβουλευτές ε, δεν εκπροσωπούν μόνο την εκλογική τους περιφέρεια, εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τη χώρα από την οποία προέρχονται. Βλέπω κάποιους ε, να γνέφουν αρνητικά, αλλά αυτό είναι και το νόημα. Εδώ νομοθετούμε για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά γνωρίζουμε τα συμφέροντα και τις νοοτροπίες ε, του τόπου από τον οποίο προερχόμαστε, αλλά ο ευρωπαϊκός νόμος είναι ευρωπαϊκός νόμος είναι νόμος όχι μόνο για τη Γερμανία, τη Γαλλία ή άλλη χώρα, είναι κοινό νόμος για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι δύσκολο για τους να το δεχτούν, αλλά εδώ και 40 χρόνια έτσι έχουν τα πράγματα. Και εάν δεν έχουν έτσι τα πράγματα, τότε ας ξεχάσουμε την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έχουμε τα Ηνωμένα Έθνη, έχουμε το Συμβούλιο της Ευρώπης, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως είναι διαφορετική. Σε ποιον άλλο να απαντήσω. Diane James, ε, ε, σε ευχαριστώ για την επικοδομητική σου παρατήρηση. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι ακόμα και η UKIP θεωρεί ότι δεν υπάρχει ε, εγγύηση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε. Α, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. δεν είσαστε πια στη UKIP. Έχετε τη δική σας άποψη. Μάλιστα, καλό αυτό. Πολύ σωστά είπατε όμως ότι χρειαζόμαστε εκλογικούς ε, καταλόγους και μάλιστα εγκαίρως ε, πριν τις εκλογές. Ε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιος έχει δικαίωμα ψήφου και το Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το κάνει πάρα πολύ καλά. Όπως ε, ήδη είπα, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η χώρα που ε, εκπονεί νωρίτερα τους ε, εκλογικούς καταλόγους και που ορίζει τους υποψήφιους. Ενώ άλλες χώρες το κάνουν αυτό πολύ λίγο πριν τις εκλογές και έτσι συμβαίνουν διάφορα λάθη. Ε, να ψηφίζει κάποιος ε, δύο φορές, για παράδειγμα, το να μην είναι γνωστό ποιος είναι καταχωρημένος ε, στη δική μου χώρα, ε, ποιος έχει διπλή υπηκότητα, διότι όταν είναι τόσο σύντομο το χρονικό διάστημα δεν υπάρχει χρόνος να γίνουν οι έλεγχοι. Βέβαια, το να ψηφίζει κανείς δύο φορές είναι καλύτερο από το να μην ψηφίσει καθόλου, αλλά σωστό δεν είναι. σύμφωνα με τους κανόνες. Θέλουμε λοιπόν ε, να γίνεται αυτό νωρίτερα, 8 εβδομάδες πριν τις εκλογές, κάποιοι θέλανε 12 εβδομάδες, αλλά ε, στις μεγάλες χώρες έχουμε εκατομμύρια πολίτες, ε, πολλούς με διπλή υπηκότητα. Θα πρέπει λοιπόν εγκαίρως να προετοιμάζονται οι εκλογικοί κατάλογοι. Ε, εκλογή μάλλον ψήφος ε, πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτες χώρες. Ε, ταξιδεύουμε πολύ. Μερικοί πρέπει για λόγου επαγγελματικού να βρίσκονται σε τρίτη χώρα κατά τον χρόνο διεξαγωγή των ευρωεκλογών. Ε, πιστεύουμε ότι είναι σωστό να συμμετέχουν οι άνθρωποι αυτοί στις ευρωεκλογέ. Τώρα, εάν κάποιος ε, μένει διαβίου σε ξένη χώρα και δεν έχει στόχο να επιστρέψει, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να το συζητήσουμε. Ε, εμείς θέλουμε να ε, προτείνουμε ψήφο στα 16. Αυτό μάλλον δεν θα συμβεί, αλλά ίσως να υπάρχει ε, κάποια σύσταση του Συμβουλίου προς τα κράτη-μέλη να εξετάσουν την πρόταση αυτή. Εγώ νομίζω ότι άνθρωποι 16 ετών είναι σε θέση να ψηφίσουν και πιστεύω ότι θα πρέπει νωρίς να τους καλούμε να συμμετάσχουν στην ε, ιστορία της Ευρωπαϊκής Συμφιλίωσης. Επίσης, όσον αφορά την ε, ηλεκτρονική ψήφο. Ε, και εδώ να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να εξετάσουμε τη δυνατότητα. Η Εστονία ήδη το εφαρμόζει αυτό, άλλοι βρίσκονται καθοδόν αφού λυθούν τα προβλήματα με την ασφάλεια των δεδομένων, ε, ίσως ε, θα ήταν χρήσιμη ιδέα. Βλέπω ότι ε, στις Ηνωμένε Πολιτείες, ε, σε τρεις πολιτείες γίνεται επανυπολογισμός των ψήφων. Είναι αδύνατον να πετύχει κανείς τα ανώτατα επίπεδα ασφαλείας. Ο συνάδελφος Μαχού από το Βέλγιο επίσης είπε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει κατόφλι σε 26 κράτη-μέλη υπάρχει τέτοιο κατόφλι. Δύο χώρες δεν έχουν, η Ισπανία και η Γερμανία. Γνωστό είναι αυτό. Και έχουν ε, λάβει έδρα στο Κοινοβούλιο άνθρωποι με το 0,7% των ε, ψήφων, ε, ενώ άλλοι χρειαζόντουσαν 700.000 ψήφους. Ίσως λοιπόν είναι απαραίτητο να καθορίσουμε ένα κατόφλι για να μπορεί να λάβει κανείς έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Σιγκόφσκι από την Πολωνία είπε ότι οι πολίτες λόγω άλλων προβλημάτων ε, δεν προσέρχονται σε ευρωεκλογέ. Οι ευρωεκλογέ ε, θα είναι πάντα πρόβλημα διότι οι Βρυξέλλες αυτομάτως ε, ούτως ή άλλως βρίσκονται πιο μακριά από ότι το Δημαρχείο της πόλης σας. Ή από ότι η πρωτεύουσα της χώρας σας με αυτό θα είμαστε για πάντα αντιμετωποί. Και στις Ηνωμένε Πολιτείες η Ουάσιγκτον ε, είναι μια εχθρική εικόνα, όπως και οι Βρυξέλλες στην Ευρώπη. Εν μέρη δικαιολογημένα, εν μέρη όχι. διότι συχνά χρησιμοποιείται και ως σκιάχτρο για να ε, ε, καλυφθούν άλλα προβλήματα για τα οποία δεν είναι υπεύθυνε οι Βρυξέλλες. Πάντα λοιπόν ε, θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα στις ευρωεκλογέ. Νομίζω ότι ε, η συνάδελφος από την ε, Καταλωνία αναφέρθηκε στο να ψηφίζουν ε, και οι άνθρωποι που βρίσκονται εντό της Ευρωπαϊκής και όχι μόνο οι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έχουμε πολλούς ε, ανθρώπους από άλλες χώρες που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σε κάποιες χώρες οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τις δημοτικές εκλογές. Έχουμε συζητήσει ήδη το θέμα αυτό, αλλά όσον αφορά τι ευρωεκλογέ δεν έχουμε προχωρήσει τόσο ακόμα. Ελπίζω λίγο πολύ να απάντησα στις ερωτήσεις σας. στον κύριο Σινόφσκι να πω ότι πάντα λέγεται ότι έχουμε δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό έχει καταλήξει να είναι σύνθημα, έχει επαναληφθεί πολλές φορές παρότι δεν ισχύει όσον αφορά το Ευρωκοινοβούλιο. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα. Ε, είμαστε αποτέλεσμα δίκαιων και ανοιχτών εκλογών όπως και η συνάδελφοι στα Εθνικά Κοινοβούλια. Έχουμε λοιπόν ε, ακριβώς ε, την ίδια νομιμοποίηση με τους βουλευτές των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων. Το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές επικύλει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος και για τις εθνικές εκλογές. Η νομιμοποίηση όμως υπάρχει. και συζητάμε ε, με εξίσου διαφανή τρόπο, πόσο μάλλον που ε, μεταδίδονται στο διαδίκτυο οι συνεταιριάσεις μας. Σε πολλά άλλα κοινοβούλια δεν συμβαίνει αυτό. Εγώ δεν αναγνωρίζω να υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι μάλλον το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να μεταφέρουμε το μήνυμά μα. Ε, δεν θα έλεγα ότι έχουμε έλλειμμα πληροφόρηση, διότι σήμερα ε, μπορεί κανεί να πληροφορεί όσο θέλει, αλλά ε, πράγματι οι Βρυξέλλε είναι πιο μακριά από τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί αποτυχία και των κομμάτων Αυτός είναι και ο λόγος που θέλουμε να επιφέρουμε κάποιες βελτιώσεις. Με το λογότυπο θέλουμε να γίνουν πιο ορατά τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Θέλουμε να υπάρχει συνεργασία εντός των πολιτικών οικογενειών και να ορίσουμε την προστιθέμενη αξία της Ευρώπης. Κυρία Χίπνερ, αυτή ήταν η απάντησή μου. Ευχαριστώ, Γιο. Θα ήθελα εν συντομία να αναφερθώ και εγώ σε κάποια από τα θέματα τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν. Καταρχάς, ε, αυτή η άποψη που εξέφρασαν ε, δύο-τρεις συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια για το κατά πόσον χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Χρειαζόμαστε για το λόγο που πολύ σαφώ εξέφρασε ο Φιλίπ Μαού. Είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και γιατί η συνθήκη διευκρινίζει σαφέστατα στο 2.3.1 ε, λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, εκπονήσει πρόταση για το σύστημα των ευρωεκλογών. Επομένως, η συνθήκη μας προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Είτε ε, να έχουμε ένα ομοιόμορφο καθεστώς ε, μεταξύ των πρωτών μελών ή να έχουμε ένα καθεστώς το οποίο βασίζεται σε κάποιες κοινέ αρχές. Το έχουμε συζητήσει και συμφωνήσαμε ότι ο καλύτερος τρόπος προκειμένου να σεβαστούμε την ποικιλομορφία, της παραδόσεις και να σεβαστούμε καλύτερα τι αρμόζει καλύτερα για τους πολίτες και σε τι είναι ε, συνηθισμένοι, ε, καλό θα ήταν να έχουμε κάποιες βασικές αρχές. Και η όλη φιλοσοφία αυτής της νομικής πράξης είναι ο σεβασμός των κοινών αρχών. Αφήνουμε μεγάλη ευελιξία στις εθνικές παραδόσεις, αν μου επιτρέπετε να τις αποκαλέσω έτσι. Και βεβαίω είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σε αυτή την νομοθετική πράξη υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτική φύσεως, αλλά υπάρχουν και αρκετές συστάσεις ε, που πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη για το μέλλον και ε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα παιδιάων ετών, 16 ετών να ψηφίσουν, κάτι το οποίο επιτρέπεται στην Αυστρία, το έχουμε βάλει για περαιτέρω προβληματισμό. Ε, είπε και η κυρία Τζέκινς και το αντιλαμβάνουμε ότι οι νέοι άνθρωποι πρέπει να αντιληφθούν ότι είναι και υποχρέωση η ψήφος. Δεν είναι απλώς η ευχαρίστηση και το δικαίωμα να αποφασίζει κάποιος, αλλά είναι και μία υποχρέωση. Επομένως, απλώς επισημαίνουμε κάποια πράγματα για το μέλλον. Δεύτερον, θα ήθελα να γνωρίζετε ότι αυτό το οποίο προτείναμε τελικά έχει προκύψει μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια για εξέβρεση συμβιβασμού. Διότι εμείς στο Κοινοβούλιο δεν έχουμε απλώς 8 διαφορετικές πολιτικές ομάδες, έχουμε περίπου 300 πολιτικό κόμματα. Έχω ξεχάσει ακριβώς ποιος είναι ο αριθμός. Προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε ένα συμβιβασμό όχι μόνο μεταξύ των πολιτικών ομάδων και των εθνικών αντιπροσωπιών, διότι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Καθήρης από εμά έρχεται και με το εθνικό του παρελθόν, ε, σε πράγματα στα οποία είναι συνηθισμένος. Και κάποιοι από τους, συνάδελφους, ε, ε, από τους συναδέλφων έχουν συμμετάσχει αρκετέ φορές στις ευρωεκλογέ και καταλαβαίνουν τι εννοείται. Αλλά για τη δημοκρατία, για να μπορέσουν οι ευρωεκλογέ να είναι πιο ίσες και να μπορούν οι πολίτες να έχουν το ίδιο δικαίωμα να γνωρίζουν ποιος θα είναι στη λίστα ε, ταυτόχρονα στο ψηφοδέλτιο. Ε, συνέβη και το εξή. Κάποιοι τρει μήνε ήδη ε, πριν από τι εκλογέ γνωρίζουν ποιον θα ψηφίσουν, γνωρίζουν και μπορούν να μελετήσουν του υποψηφίου και στι τελευταίε εκλογέ είχαμε και περιπτώσει τι οποίε δύο εβδομάδε πριν από τι ευρωεκλογέ δεν υπήρχε ψηφοδέλτιο. Επομένω, ε, γι' αυτό ακριβώ προτείνουμε και την εναρμόνιση ε, και τι συγκεκριμένε προθεσμίε για την εκλογική διαδικασία δεν ε, είναι και κάτι όμως ε, το οποίο είναι ε, και υποχρεωτικό να το κάνουμε. Αναζητούμε εδώ ένα συμβιβασμό που θα επιτρέψει σε όλους να νιώσουν ικανοποιημένοι. Και θα ήθελα επίσης να τονίσω αυτό το οποίο κάνετε κι εσείς άλλωστε, και συνάδελφοι, δεν θεωρούμε ότι μέσω του συστήματος των εκλογών αυτομάτως ε, θα προκύψει ε, μεγάλη συμμετοχή. Εάν όμως ο κόσμος διαπιστώσει ότι η εκλογική διαδικασία τους δίνει περισσότερες πληροφορίες, τους προσφέρει και το δικαίωμα να έρθουν σε επαφή με τον άνθρωπο που θα εκλεγεί, να γνωρίσουν κάποια περισσότερα πράγματα για αυτό, να γνωρίζουν επακριβώς τι θα κάνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε ποια πολιτική ομάδα θα είναι, ε, τι πολιτικό πρόγραμμα θα έχει ομάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι δημοκρατία. Να ε, αναζητήσουμε την αλήθεια, τα γεγονότα. Κάτι το οποίο φαίνεται να αγνοούμε στις ε, πολιτικές διαδικασίες. Ε, μας ενδιαφέρει λοιπόν η ισότητα των πολιτών και οι χρηστές δημοκρατικές πρακτικές και η ποιότητα της δημοκρατίας. Για κάποια συγκεκριμένα πράγματα τώρα. Ο νόμος αυτός ελπίζουμε ότι θα ε, προκύψει φέτος. Φέτος ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και τη διαδικασία του Brexit. Δεν ξέρουμε πότε ε, και αν θα υπάρξει, αλλά λαμβάνουμε υπόψη και το θέμα της κατανομής των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και επομένως πρέπει να το κάνουμε. Υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πρέπει να γίνει ε, τώρα αυτό, να μην καθυστερήσει. Και φυσικά η συζήτηση για τον εκλογικό νόμο γίνεται και μεγαλύτερη πρόκληση. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε και περιμένουμε και συζητήσεις στα Εθνικά Κοινοβούλια όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία της κύρωσης εμείς ως ε, βουλευτές που εκπροσωπούμε πολίτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο είμαστε διατεθειμένοι να ε, δούμε το θέμα αυτό του μελλοντικού κοινοβουλίου, τις διαφορετικές προοπτικές, να λάβουμε υπόψη μας όλες τις προκλήσεις και την κατανομή των εδρών και την πολιτική απόφαση για το πώς ε, θα υλοποιηθούν όλα αυτά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, αυτό είναι το τελευταίο που θα ήθελα να κάνω. Δεν υποχρεώνουμε αλλά προτείνουμε μια προσέγγιση. Και αυτό φαίνεται από την ημερομηνία των εκλογών, διότι υπάρχουν διαφορετικέ παραδόσει. Άλλοι ψηφίζουν Πέμπτη, άλλοι ψηφίζουν Παρασκευή, άλλοι Σάββατο, άλλοι Κυριακή. Ουσιαστικά έχουμε μια εβδομάδα ευρωεκλογών και αυτό δεν θέλουμε να τα αλλάξουμε. Δεν προτείνουμε μία μέρα για όλου. Πιστεύουμε όμω ότι πρέπει να σταματήσουν αυτέ οι τέσσερι ημέρε εκλογή των υποψηφίων την ίδια ημέρα. Εκεί προτείνουμε μια κάποια εναρμόνιση δηλαδή. Το βράδυ της Κυριακής ε, να ολοκληρώνονται όλες οι εκλογικές διαδικασίες και να υπάρχει μια μεγάλη ευρωπαϊκή εκδήλωση με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών ταυτόχρονα. Αυτό ε, θέλουμε. Τέτοιας μορφής εναρμόνιση προτείνεται σε αυτή την περίπτωση. Και κάτι τελευταίο για τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου υποψήφιο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Spitzenkandidat. Ε, είναι ένα ζήτημα το οποίο ε, είναι δύσκολο όταν το συζητούμε με το Συμβούλιο και κυρίως καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι νομικά η στιγμή για αυτή την ε, λύση. Αλλά αν δείτε τι γίνεται στα ευρωπαϊκά κόμματα και στις ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες, οι περισσότεροι εξ αυτών, τουλάχιστον τα μεγάλα πολιτικά κόμματα, τέτοια προσέγγιση ακολουθούν στο καταστατικό τους. Επομένως, ε, πολιτικά ισχύει αυτό στην Ευρώπη. Μπορεί να μην ε, εγγράφεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και στο, νομοθεσία, στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά δεν μπορούμε να αποφύγουμε και τις εξελίξεις, γιατί από ό,τι φαίνεται τα πολιτικό κόμματα αυτό επιθυμούν. Δεν μπορούμε λοιπόν να κοφεύουμε, διότι αυτά προκύπτουν από πολιτικά θέλω, από πολιτικά ε, πολιτικές παραδόσεις και ε, αυτό σημαίνει ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και έτσι κινούμαστε μέσω μιας ε, αμυγούς δημοκρατικής διαδικασίας και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση που απορρέουν από τη συνθήκη αλλά θέλουμε αυτό να γίνει από κοινού με τους συναδέλφους μας σε εθνικό επίπεδο και με τις κυβερνήσεις διότι θεωρούμε ότι αποτελεί κοινή πρόκληση και κοινή ευθύνη. Μπορεί βέβαια κάποια πράγματα μετά από τη σημερινή συζήτηση να τερμινεύεται διαφορετικά. Πραγματικά θα ήθελα να σας ζητήσω να λάβετε υπόψη ε, ε, το θέμα ως κοινή πρόκληση, να μην ε, αγνοήσετε τη δημοκρατική διαδικασία και τις εκλογές, αλλά να κάνουμε ένα βήμα προς την αξιοπιστία αυτή τη διαδικασία ή τουλάχιστον αυτό θεωρούμε εμείς και προς την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Αυτό είναι το διακύβευμα ε, κατά την άποψή μου. Θα ολοκληρώσουμε λοιπόν με αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη που σημαίνει ότι έχετε λίγο χρόνο να διασκεδάσετε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, το γεύμα είναι στο Ισόγειο, ε, στο εστιατόριο στη μία η ώρα. Να σας ε, καλέσω λοιπόν καταρχάς το γεύμα και μετά θα συναντηθούμε στις 3 για να συζητήσουμε την αλλαγή της Ευρώπης, τις μελλοντικές συνθήκες και την εφαρμογή των συνθήκων αυτή τη στιγμή.